meeting. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ας ξεκινήσουμε μόλις ε, καθίσουν όλοι. Σας καλωσορίζω μετά τις ε, καλοκαιρινές διακοπές του συναδέλφου, τα μέλη, τη γραμματεία, όλους. Και ελπίζω να συνεχίσουμε με μια φιλική ατμόσφαιρα στην Επιτροπή μας για να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πολίτες που έχουν στραφεί προς εμάς. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω ενστάσεις. Τα πρακτικά της συνεδρίας του Ιουνίου, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Έχω μερικές ανακοινώσεις σήμερα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα στις 2.30 ε, θα κάνουμε μια κοινή συνειδρίαση με την ΑΦΚΟ για την ειδική έκθεση του δημοσιο... της Δημοσιολαβήτριας για τη διαφάνεια στο Συμβούλιο. Θα διαρκέσει 45 λεπτά και μετά θα συνεχίσουμε με τις κανονικές μας εργασίες. Πάμε στο επόμενο τμήμα. Διάφορες αλλαγές στη γραμματεία που έγιναν το καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα η κυρία Σιλβί Ρένερ που εργάστηκε ως βοηθός στη ΣΠΕΤΗ για 13 χρόνια συνταξιοδοτήθηκε στα τέλη Αυγούστου. Η Σιλβή ήταν μία από τις συναδέλφους που είχε άμεσες επαφές με τους αναφέροντες όταν έρχονταν στις συνεδριάσεις μας. Ε, είχε ασχοληθεί με την αλληλογραφία και πολλά άλλα καθήκοντα είχε αναλάβει στη γραμματεία και ήθελα να την ευχαριστήσω. Δεν βρίσκεται εδώ να την ευχαριστήσω για τον επαγγελματισμό της, την ευγένειά της και τις προσπάθειές της. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά ίσως να μας παρακολουθεί από το διαδίκτυο. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι η Φάνη Φοντέν, επίσης ε, διοικητικό προσωπικό, ε, μετατέθηκε στη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και της εύχομαι πολύ καλή τύχη σε αυτή την επιτροπή και με μεγάλη μας ε, δεν μας πήραν μόνο μέλη της γραμματείας φέτος το καλοκαίρι. Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοίνω ότι η Πατρίσια Βαντεπέρ, μια ε, πολύ ε, έμπειρη ε, νομικός ε, και υπάλληλο που εργάστηκε για πολλά χρόνια στη Λίμπε και πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Πρεσία Υποστήριξη του Ασύλου στη Μάλτα, αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί μας από σήμερα. Πατρίσια, δείξτε, σηκώστε το χέρι να συστηθείτε. Και τον Ιούλιο επίσης λάβαμε και μια ενίσχυση από την Ισπανία, τον Χεσούς Ράμος Καρσία, που θα εργαστεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ως εθνικός εμπειρογνώμων στη γραμματεία μας. Έχετε μεγάλη σταδιοδρομία στην ε, διοίκηση στην Ισπανία και εσείς πείτε μας ποιος είστε, ορίστε, καλώς ορίσατε. Και τέλος, η ομάδα έχει μια νέα βοηθό, την Κριστίνα Κόβατς είναι από την Ουγγαρία, έχει εργαστεί σε διάφορα τμήματα της Κομισιόν και πριν πολύ καιρό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι πριν πολύ καιρό, είναι ακόμα νέα. Ορίστε και εσείς καλώς ορίσατε όλοι. Με μεγάλη μας χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας. Και σας λέω προσωπικά, αν κάποιος δεν σας συμπεριφέρεται καλά, να με πάρετε τηλέφωνο. Δεν έχουμε άλλα ε, στο σημείο 5 εκτός από ένα θέμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Αφορά τον κανονισμό για τον οποίο η συγγήτρια η κυρία Βαλέντσα είπε ότι αποσύρεται ως η συγγήτρια και τώρα μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Το ΕΛΚΑ τον αντικατέστησε γρήγορα και έτσι ο κύριος Πρέντα διορίστηκε ως εισηγητής. Θα αναλάβει λοιπόν καθήκοντα την επόμενη εβδομάδα. Όσον αφορά την ε, συμπεράσματα της συνεδρίας των συντονιστών, πρώτα απ' όλα ε, εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη του Οκτωβρίου και συμπεριλάβαμε τις ε, αναφορές 0825, 0963, και συμπεριλάβουμε και τι επίσης τις 0189, 0250, 0328 στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε και μία συνεδρίαση με την Επιτροπή Αναφορών του Bundestag, όπως είπαμε, όσον αφορά τις προσβαλόμενες συστάσεις. Οι ε, συμβιβαστικέ προτάσει εγκρίθηκαν σε πολλέ περιπτώσει εκτό από την αναφορά 0313 που θα διατηρηθεί ανοιχτή και θα σταλεί επιστολή στι Ισπανικέ Αρχέ και την αναφορά 0317 που θα κλείσει. Η 0318 δηλώθηκε παραδεκτή και έκλεισε. Και πέραν αυτών οι συστάσεις μου εγκρίθηκαν. Για τα σημεία Β μια λεπτομερής λίστα των αποφάσεων θα συμπεριληφθεί στα γραπτά συμπεράσματα όσον αφορά τι διερευνητικέ αποστολέ και ακρόασει. Πρώτα απ' όλα η επίσκεψη συντονιάνα τη Ισπανία, οι συντονιστές σημείωσαν το, τελικό πρόγραμμα της αποστολή και την τροποποιημένη λίστα συμμετοχόντων συμπεριλαμβανομένη τη συμμετοχή τεσσάρων μέλων οφήσιο. Για την επίσκεψη στη Βαλεντόρα στην Ιταλία τον Οκτώβριο, μετά από μια μεγάλη ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκε να διερευνήσουμε περαιτέρω σε ποια ημερομηνία θα γίνει η διερευνητική αποστολή. Η γραμματεία θα την κοινοποιήσει μέσω επικοινωνίας με τους συναδέλφους με γραπτή διαδικασία. Η ακρόαση για τα άτομα με αναπηρία εγκρίναμε το προσωρινό πρόγραμμα το οποίο θα λάβει η χώρα 9 Οκτωβρίου. Ε, θα σας στείλει την τελική έκδοση η γραμματεία και η προετοιμασία για τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια στις 27 Νοεμβρίου. Επίσης συζητήθηκε ενημερωτικά ε, θέματα, τα σημείωσαν οι συντονιστές και δεν υπήρχε τίποτα υπό τα διάφορα. Αυτά για τους συντονιστές ως και τις αποφάσεις τους. Κύριε Τερικάμπρας, Συγγνώμη, αναφέρατε ότι ο κύριος Βαρέσα χρειάστηκε να αντικατασταθεί ως εισηγητής. Ελπίζω να γίνει αυτό στη συνεδρία των συντονιστών, διότι αυτή είναι η μέθοδος. Αυτή είναι η διαδικασία. Ήταν και δύσκολη απόφαση στη συνεδρία των συντονιστών που τον διόρισε ο συντονιστής. Πρόεδρος, ναι, αλλά ξέρετε τι, αυτό δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Διότι το ΕΛΚ έχει αυτή τη θέση την οποία αγοράσαν με πόντους παλαιότερα. Και το ΕΛΚ λοιπόν έχει την ελευθερία να επιλέξει να αντικαταστήσει τον κύριο Βαλέσσα με όποιον θέλει. Δεν είναι διορισμός σαν τους άλλους, διορισμός γιατί όπως κάνουμε βάσει πόντων κτλ. Και, και της ε, σχετικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει τώρα διότι ο κύριος Βαλέσσα αποσύρεται διότι θα θέσει υποψηφιότητα ως δήμαρχος της πόλης του Γκτάνσκ οπότε χρειαζόμαστε μια γρήγορη απόφαση και ο κανόνας λέει ότι πρόκειται για έδρα του ΕΛΚ και το ΕΛΚ μπορεί να επιλέξει όποιον θέλει προς κατάσταση του εισηγητή. Το συγγνώμη, αλλά έτσι έχει διαδικασία. Να προχωρήσουμε. Πάμε στην αναφορά 48 για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην πόλη της Βαλένθια. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον, αλλά έχει στείλει δύο έγγραφα με 800 επιπλέον υπογραφές, που είναι πολλές. Εκπρόσωπος της Κομισιόν εδώ. Σας παρακαλώ πάρτε το λόγο να μας διαφωτίσετε για την αναφορά αυτή. Muchas gracias, señor presidente. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για το γεγονό ότι οι τοπικές αρχές της πόλης της Βαλένθια τροποποίησαν την κυκλοφορία και έτσι μία λεωφόρος της πόλης που ήταν μονόδρομος έγινε τώρα διπλής κατεύθυνσης. Ως συνέπεια οι αναφέροντες καταγγέλουν ότι τα επίπεδα ε, της κυκλοφορίας αυξήθηκαν πολύ, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα και αύξηση των εκπομπών ρηπογόνων ουσιών. Υπάρχει μεγαλύτερη χορύπαυση επίσης και έτσι πλήττεται η ποιότητα της ζωής των γειτόνων. Ζητούν λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσουν από τις Ισπανικές Αρχές να τροποποιήσουν αυτό, αυτή την κυκλοφοριακή ρύθμιση και έτσι η λεωφόρος αυτή η Ντελοέστε της Ανατολής στη Βαλένθια να γίνει και πάλι ε, μονής κατεύθυνσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ πρέπει να πει, όπως το κάνει πάντα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει μόνο στις υποθέσεις εκείνες που καλύπτονται από το κοινοτικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ρύθμιση κυκλοφοριακή σε τοπικό επίπεδο δεν ρυθμίζεται από το ενωσιακό δίκαιο. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των χωρών μελών. Ε, αυτό βέβαια δεν σημαίνει από την άλλη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει και δεν οφείλει να ελέγχει τα επίπεδα ρήπανση στο περιβάλλον εξαιτία τη κυκλοφορία. Ε, πρέπει να εξετάζει την ποιότητα του αέρα και την ρήπανση του αέρα. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει συστηματικά την τήρηση από πλευρά των χωρών μελών των οριακών τιμών για όλες τις ρηπογόνες ουσίες ή τα σωματίδια. Και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή συγκεκριμένη η ευρωπαικη εξετάζει να δει κατά πόσο η συγκέντρωση τέτοιων ρηπογόνων ουσιών είναι ή όχι πάνω από τις οριακές τιμές στις διάφορες ζώνες, πόλεις κλπ. Για το κυκλοφοριακό οι ρηπογόνες ουσίες, οι πιο ανησυχητικές, είναι το διοξίδιο του αζότου και τα σωματίδια, το PM10. Για αυτές τις δύο ουσίες λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις εκθέσεις ποιότητας ε, που εκδίδει η Ισπανική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και διαπίστωσε ότι όσον αφορά την περιοχή της Βαλένθια δεν έχουν καταγραφεί τιμές πάνω από τις οριακές τιμές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει παράβαση της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή της Βαλένθια. Όσον αφορά την ηχορύπανση, η οδηγία για την ηχορύπανση απαιτούν από τις χώρες μέλη να προσαρμόζουν παντού κάποιους χάρτες ηχορύπανσης έτσι ώστε να ξέρουμε ότι δεν πλήττεται η υγεία των πολιτών από υπερβολική χορύπανση. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκίνησε διαδικασίες κατά παραβάση σε βάρος των χωρών εκείνων που δεν έχουν εγκρίνει ακόμα τέτοια έγγραφα έτσι όπως προβλέπει η οδηγία. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία και έτσι η διαδικασία αυτή ακολουθεί το δρόμο της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει καταλήξει τη λύση, δεν το έχει λύσει δηλαδή το ζήτημα. Να ξέρετε ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να ενημερώνει την Επιτροπή σας για την συνεχιζόμενη αυτή διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Οι Ευρωβουλευτές τώρα έχουν το λόγο. Ρώσα. Πρώτον, θα μπορούσαμε να είχαμε ε, συνδέσει την ε, αναφορά αυτή με άλλη αντίστοιχη για τη Μαδρίτη. Αναβλήθηκε όμως γιατί δεν μπορεί να είναι εδώ αναφέρον. Ούτε και εδώ όμως είναι οι αναφέροντες παρόντες, οπότε δεν βλέπω γιατί αναβάλαμε αυτή για τη Μαδρίτη για άλλη εβδομάδα ενώ εξετάζουμε αυτή για τη Βαλένθια. Υπάρχει εξάλλου και μελέτη που έχουμε αναθέσει εμείς οι ίδιοι για την ρήπανση του αέρα. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί αναβλήθηκε αυτή για την ε, Μαδρίτη, ενώ κάνουμε τη συζήτηση και εξετάζουμε την αναφορά αυτή για τη Βαλένθια. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα. Διάβασα τι λένε οι αναφέροντες. Τώρα πέρα από την ηχορύπανση αυτή και την ατμοσφαιρική ρήπανση, αυτό το οποίο παρουσιάζουν στα έγγραφά τους και λένε είναι ότι δεν υπάρχουν οι ανοιχτευτές συγχωρήπανσεις εκεί που θα έπρεπε. Αλλά σε άλλα σημεία μακριά. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κανείς είτε την ηχορύπανση είτε ακόμα και την ε, ατμοσφαιρική ρύπανση, γιατί και αυτοί οι ανιχνευτές βρίσκονται μακριά από το κέντρο. Έχουν μπει ανιχνευτές, έτσι λένε τουλάχιστον οι αναφέροντες, μακριά στην άκρη της πόλης, άρα τα στοιχεία τα οποία ε, συσσωρεύονται με τον τρόπο αυτό δεν είναι αξιόπιστα. Η πρότασή μου είναι η εξή. Δεδομένου ότι η Κομισιόν είπε ότι όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση, τα στοιχεία, λέει, η Κομισιόν είναι εντάξει, αλλά αναφέρον λέει ότι δεν είναι, γιατί ακριβώ οι ανιχνευτέ βρίσκονται μακριά από το κέντρο. Και επίση η Κομισιόν είπε ότι για την ηχορύπανση υπάρχει ανοιχτή διαδικασία να παραμείνει λοιπόν ανοιχτή η αναφορά αυτή, να σταλεί επιστολή στον Δήμο της Βαλένθιας, αρχές της πόλης, ώστε να μας εξηγήσουν τι πιστεύουν για αυτό το θέμα και να πάει η υπόθεση αυτή και στην Επιτροπή ΕΝΒΗ, ώστε και εκείνη να αξιολογήσουν λίγο το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και να συνεχιστεί βέβαια η επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μας ενημερώνει και για τη διαδικασία επιπαραβάση, για την ηχορύπανση, αλλά να ψάξουν να βρουν πού βρίσκονται αυτοί οι ανιχνευτές για να ξέρουμε είναι εξόπιστα τα στοιχεία που έχουμε ή όχι, να δούμε τελικά ποιο έχει δίκιο, αναφέρον ή όχι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριο Μαρσελέση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ με προσοχή μελέτησα την αναφορά, άκουσα και όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευχαριστώ γιατί συμφωνώ με πολλά που είπε. Όντω, για να καταλάβουμε την υπόθεση αυτή καλά, πρέπει να θυμηθούμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ενέκρινε ένα σχέδιο ε, βιωσιμότητας και για την ε, Βαλένθια, αλλά δεν άρχισε να ισχύει. Και η νέα αυτή κυβέρνηση, που είναι λίγο καιρό τώρα, έχει αρχίσει την εφαρμογή αυτού του προγράμματος βιωσιμότητας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και μέτρα για την ατμοσφαιρική ρήπανση, για το κυκλοφοριακό. Ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη πόλη Βαλένθια και το κυκλοφοριακό είναι πολύ σημαντικό για την υγεία. Στα διάφορα μέτρα λοιπόν που προβλέπονται, προβλέπεται να αλλάξει και η κυκλοφοριακή ρύθμιση στη λεωφόρο αυτή, που ήταν ε, ε, μονής κατεύθυνσης και τώρα έγινε διπλής. Από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 φαίνεται ότι τα πράγματα πήγανε καλά. Η αλλαγή αυτή που έγινε μείωσε από ό,τι φαίνεται την ένταση ε, της κυκλοφορίας. Από 12.000 οχήματα πήγανε σε 10.000. Άρα 23% μειώθηκε το κυκλοφοριακό, κάτι το οποίο επέτρεψε να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και αυτό το λένε όλες οι μετρήσεις. Το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναγνωρίζει επίσης ότι βελτιώθηκε και το θέμα της συγχωρήπανσης και επιπλέον έχουν ληφθεί και άλλα μέτρα όπως είναι η έγκριση μιας ε, διαδικασίας για τη μέτρηση του αέρα, λαμβάνονται στοιχεία και σε σχολεία και σε γυμνάσια και υπάρχουν και νέες εγκαταστάσεις μέτρησης. Οπότε η αλλαγή είναι αρκετά δραστική τα τελευταία, ε, τους τελευταίους μήνες και έχουμε επιτέλους καλές μετρήσεις, σωστές, έχουμε ένα συνολικό σχέδιο και νούμερα, το οποίο, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνονται καλά. Οπότε θα πρότεινα να κλείσει η αναφορά αυτή, γιατί είδαμε ξεκάθαρο ότι υπάρχει ουσιαστική βελτίωση. Και επιπλέον, μην αφήνουμε τέτοιες ε, αναφορές να μας κάνουν να παρεμβαίνουμε σε τοπικά ζητήματα όπως αυτό που είναι πολύ τοπικό στη Βαλένθια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τερικάμπρας. Ευχαριστώ. Τα στοιχεία... Τα στοιχεία που ακούσαμε, όπως είπε ο κύριος Μαρσελέση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κάνουν να καταλήξω στο εξή. Λέτε, δεν υπάρχει ατμοσφαιρική ρήπανση. Η χορύπανση φαίνεται ότι υπάρχει. Υπάρχει στο συγκεκριμένο δρόμο για τον οποίο μιλάει ο αναφέρον. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Έτσι μιλάει για ένα συγκεκριμένο δρόμο, μια συγκεκριμένη λεωφόρο. Τώρα, εμένα πραγματικά με προβληματίζει πραγματικά πολύ. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αυτή πρέπει να ασχοληθεί με την κυκλοφορία σε ένα δρόμο μίας πόλης της Ισπανίας. Μα να αρχίσουμε έτσι. Αν μας πούνε Μα το πεζοδρόμιο ή το δόστρωμα ή τα παιδιά τελικά παίζουν μπάλα στο δρόμο και σπάνε τζάμια, δεν σπάνε κτλ. Αν αρχίσουμε να ασχολιόμαστε με τέτοια συγκεκριμένα ζητήματα, ε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Φοβάμαι ότι κάποια μέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εμφανιστεί γελία και άσχετη με την ουσία. Κάτι το οποίο θα ήταν κρίμα. Λοιπόν, η Επιτροπή μας πρέπει να ζυγίζει καλά τα πράγματα και να ξέρει τι ακριβώς κάνει και δεν μπορεί να ασχολείται με το τι συμβαίνει σε κάθε δρόμο της Ευρώπης. Ο αναφέρον πρέπει να αναφέρεται στο Δήμο του, να λύνει τα προβλήματα. Όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Είναι απίστευτο που συμμετέχω σε μια τέτοια συζήτηση και μετά θα μου στήσετε και να ψηφίσω. Εγώ λέω να κλείσει. Με πέντε χέρια το ζητάω αυτό. Ευχαριστώ. να παρακαλέσω τους ε, πολιτικούς σύμβουλους να μην γελάνε δυνατά τη στιγμή που μιλούν οι ευρωβουλευτές. Μετρήσει ζήτησε το λόγο, όχι η Ρώσα. Sí, Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση πολιτική εδώ στην Επιτροπή μας. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Οι δύο συνάδελφοι προτείνουν να κλείσει. Εγώ όχι. Ε, είναι θέμα πολιτικό. Επειδή είσαστε από την αριστερά και έχει η αριστερή κυβέρνηση, λέτε αυτό. Διαφωνώ. Και αφήστε με να τελειώσω. Λοιπόν, η οδηγία για την ε, ατμοσφαιρική ρήπανση και για την ηχορύπανση είναι πράγματα απολύτω αντικειμενικά. Δεν μπορεί να λέτε ότι δεν είναι ρεαλιστικά. Για μένα η αναφορά στέκει γιατί μιλάει για το περιβάλλον. Και να αναφέρον ότι οι ανιχνευτές και ο αναφέρον είναι πάντα ο πρωταγωνιστής εδώ στην Επιτροπή μας. Λέει ότι οι μετρητές βρίσκονται σε ακατάλληλα σημεία. Σε σημεία όπου δεν μπορούν να μετρηθούν τα πράγματα που θέλουμε να μετρήσουμε. Θα έπρεπε οι μετρητές να βρίσκονται στον αστικό χώρο για να μετρήσουν αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε. Λοιπόν, να ζητήσει η Κομισιόν από το Δήμο της Βαλένθια να διευκρινίσει το θέμα αυτό των μετρητών. Πού βρίσκονται για να ξέρουμε κατά πόσο είναι καλά τοποθετημένοι ή δεν είναι. Εδώ μας λέει ο αναφέρον ότι υπάρχει στο Πολυτεχνείο, σε μια άλλη ζώνη που είναι περιορισμένη στην κυκλοφορία. Ε, αν οι μετρητές δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι, πώς θα μετρήσουν την ατμοσφαιρική ρήπανση. Όλα μπορεί να είναι υπέροχα, αλλά ο αναφέρον λέει ότι οι μετρητές δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να βρεθούν. Συνεπώς, να σεβαστούμε τον αναφέροντα όπως κάνουμε πάντα η γνώμη μου είναι να παραμείνει ανοιχτή και να στείλουμε απάντηση στον αναφέροντα να πει πού βρίσκονται ακριβώς οι μετρητές και η Κομισιό να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Και μετά θα αποφασίσουμε. Αλλά μην ε, παρατάμε τον αναφέροντα έτσι. Λοιπόν, ανοιχτή. Να μην είναι ανοιχτή και εγώ με 15 χέρια. Ωραία. Eh, δεν ήθελα πριν να πάρω το λόγο, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση κάπως ιδιαίτερη. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Πάντως, στα πλαίσια αυτά, εκ μέρους της ομάδας μου, θα έλεγα και εγώ ότι επειδή δεν υπάρχει σαφήνεια για αυτή την υπόθεση, προτείνω να μην είναι ανοιχτή η αναφορά και να μας δοθεί ευκαιρία να διευκρινίσουμε όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε τώρα. Και τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Να παραμείνει ανοιχτή λοιπόν. Αυτό προτείνω. Ο κύριος Μαρσελέση. Ναι, συμφωνώ με την κυρία Εστέρας ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε τη συζήτηση. Εγώ έδωσα στοιχεία. Την πολιτικοποίηση εκείνη την έκανε. Οπότε, θα έλεγα, όπως έλεγε και ο συνάδελφος Τερικάμπρες, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η Επιτροπή Αναφορών για να γίνονται εδώ ακριβώς τέτοιοι μεροληπτικοί τσακωμοί ιδεολογικοί. Εγώ λέω ότι τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα που δίνουν εμπειρογνώμονες, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχουμε. Γι' αυτό προτείνω να κλείσει αυτή η αναφορά και ελπίζω όντω να κλείσει. Τον κάνει καλά ένας Δήμος τη δουλειά του, αυτό πρέπει να τον αγνωρίζει η Επιτροπή μας. Και αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεγάλοι δήμοι επιτέλους τώρα με την νέα κυβέρνηση άρχισαν να εφαρμόζουν προγράμματα και μέτρα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Αυτά τα σχέδια λοιπόν τώρα που εφαρμόζονται και που είναι καλά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε ότι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πολύ ωραία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλετε να προσθέσετε κάτι, να ξεκαθαρίσετε κάτι τώρα που ακούσατε τους ευρωβουλευτές. Όχι. Ωραία. Προσπαθώ να μετρήσω. Δεν έχουμε απαρτία, δεν μπορούμε καν να ψηφίσουμε. Ακούσαμε ευρωβουλευτέ που θέλουν να κλείσει, άλλοι που θέλουν να μείνει ανοιχτή. Δεν έχουμε όμω απαρτία. Δεν έχουμε τουλάχιστον 12 μέλη, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάει στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Συμφωνείτε? Εάν θέλετε οπωσδήποτε να προχωρήσει προς μια κατεύθυνση αναφορά, θα πρέπει να είναι παρόντε οι συναδελφοί σα. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ρώσα, θες κάτι να προσθέσει. Συμφωνώ απόλυτα με την Πρόεδρο και για άλλη μια φορά. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής μας αναφορών που εξετάζει τις ε, αιτήσει των πολιτών και να μην είμαστε παρόντες. Η Ρώσα το λέει ήπια. Εγώ θα το πω με πιο σκληρά λόγια. Είναι σπατάλι του χρόνου όλων και δεν είναι και θετικό απέναντι στους άλλους αναφέροντες που πιθανότατα να θέλαν να βρεθεί η δική τους αναφορά στην ημερήσια διάταξη. Όπω ε, και να έχει, μεταφέρουμε το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Με μεγάλη μας λύπη. Το 8 έχει αναβληθεί και προχωράμε στο υπαριθμό 9, τρεις αναφορές, 4, 5, 6, 3, 0, και 4, ε, και 7, 4, 0. αφορούν την Βενεζουέλα. Οι αναφέροντες είναι παρόντες και σας καλωσορίζω στην ε, Επιτροπή των Αναφορών Ιγνάσιο Φερνάντες, Πατρίσια Καρέρα Ρόχα και σας δίνω το λόγο για το πολύ πέντε λεπτά στον καθένα. Ας ξεκινήσουμε από την κυρία λοιπόν, παρακαλώ. Πέντε λεπτά ο καθένας ή πέντε λεπτά συνολικά. Ο καθένας. Ωραία, ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Έγραψα στα ισπανικά την αναφορά μου, οπότε θα μιλήσω ισπανικά. Οι σχέσεις της Βενεζουέλας ε, και της Ευρώπης ήταν πολύ στενή ήδη τον 20ο ε, αιώνα. Τις δεκαετίας του 40 και του 70 η Βενεζουέλα υποδέχτηκε πολλούς, ε, όπως και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, πολλούς, πολλά παιδιά της Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτοκαλίας, της Γαλλίας, Ελλάδας, Γερμανίας και της Κροατίας. Και υπάρχει και το έγγραφο για τη στρατηγική για τη Βενεζουέλα το 2007-2013, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει το ενδιαφέρον της και τη δέσμευσή της να βοηθήσει την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Οι σχέσεις και η βοήθεια συνεργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ξεκινήσει σε περιφερειακό επίπεδο. Η 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει από την Βενεζουέλα και όλο και περισσότεροι φεύγουν από τη Βενεζουέλα. Και ο ΙΕ πιστεύει ότι η μεταναστευτική κρίση της Βενεζουέλας είναι αντίστοιχη εκείνης της Μεσογείου. Ζούμε μια εποχή μεγάλων και γρήγορων αλλαγών. Πολλά γεγονότα λαμβάνουν χώρε σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει μια κρίση ταυτότητα πολύ ισχυρή, περισσότερο από ποτέ, που οδηγεί σε πολλές ε, πολιτικές διαφορές και σε μια ανθρωπιστική κρίση των γειτονικών χωρών πιέζει την ε, ενότητά της. Οι ψεύτικες πληροφορίες, οι μονομερείς, οι στρεβλώσεις, η μεροληψία επηρεάζουν σε όλο τον κόσμο τα, τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Βενεζουέλα είχε αποφασίσει ποιοι είναι οι φίλοι της, κάτι όμως το οποίο αλλάζει τώρα. Υπάρχουν ε, νέε ευκαιρίε βέβαια μετά από κάθε κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίε όπω είναι η ανθρώπινη εξωπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, ε, κράτο δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη πρέπει να πάρει ένα σημαντικό ρόλο υπέρ τη στήριξη των δημοκρατιών και να ζητήσει μηδέν ανοχή στην διαφθορά και στην ατιμορρησία, κάτι το οποίο θα βοηθούσε την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ηγετικό της ρόλο. Η περίπτωση της Βενεζουέλας είναι μια περίπτωση όπου χρειάζεται κάτι παραπάνω από κυρώσεις από τις παγκόσμιες κυβερνήσεις. Όπω λέει και το εγγραφο στρατηγικη στρατηγικής 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει το διάλογο με τη Βενεζουέλα, ακούγοντα ε, ε, πολλέ ε, απόψει από όλου του Βενεζουελάνου. Να στηριχτούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, όπω είναι ο Ερυθρό Σταυρό, και να βοηθηθεί ο τη της Βενεζουέλας όσον αφορά την υγεία του και την πρόσβαση σε βασικέ υπηρεσίε. Να συνεχίσει το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιών ε, όσων έχουν ανακατευτεί με την μείωση της δημοκρατία στη Βενεζουέλα και να συνεχιστεί η δήλωση ότι πρόκειται για persona non grata ε, για όσους ε, όντω συμπεριφέρονται κατά τη δημοκρατίας στη Βενεζουέλα. Εγώ είμαι και Ισπανός και Βενεζουελάνος και Ευρωπαίος και έτσι νιώθω και έτσι ταυτίζομαι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να φροντίσει τους Βενεζουλάνους και τα παιδιά της Ευρώπης στην Βενεζουέλα είναι ζωτική σημασία για να επανέλθουν οι αναγκαίε συνθήκε και οι προποθέσει για μια ευημερούσα χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας διαβεβαιώ ότι πολύ σπάνια έχουμε αναφέροντε που περιορίζονται στο χρόνο ομιλία που τους δίνουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη συνέπειά σας. Δίνω το λόγο στη συναδελφό σα. Ευχαριστώ πολύ. Με Πατρίθια Καρέρα. Και εγώ από τη Βενεζουέλα που ανησυχώ πάρα πολύ για τους θανάτους, τους βίες, όλα και από τις ασθένειες. Ε, ζητούσα την προηγούμενη εβδομάδα από τους πολίτες του κόσμου να με βοηθήσουν υπέρ των ατομικών ελευθεριών των αδερφών μας στη Βενεζουέλα. Εμείς κάνουμε κάτι που ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα κάναμε. Να έρθουμε εδώ και να μιλήσουμε για ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Είναι κάτι που πραγματικά ποτέ δεν θα φανταζόταν κανείς. Ζούμε κάτω από ένα καθεστώς, το οποίο κυριαρχού το λαθρεμπόριο, ε, πετρελαίου, όπλων. Αυτό που ενδιαφέρει όμως του, το λαό είναι να μην μας βλέπουν σαν σταγόνα πετρελαίου. Ζούμε όμως τη χειρότερη κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ <clears throat> στη χώρα μας. Χωρίς δημοκρατία, χωρίς φαγητό, χωρίς φάρμακα, χωρίς ασφάλεια, χωρίς υγεία, χωρίς αξιοπρέπεια και κυρίως χωρίς ελευθερίες. Εμείς ε, δεν ε, θέλουμε να σας ε, κουράσουμε, αλλά το να είναι κανείς πολίτης είναι ένα δικαίωμα και δεν μπορεί να χαίρει το δικαιώματο αυτού χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς <clears throat> είμαστε άνθρωποι και εμείς φτιάχνουμε τη χώρα, όχι η χώρα μας. Οπότε εμείς θέλουμε δικαιοσύνη και να μην επιτρέπονται αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γι' αυτό θέλουμε να ισχύσει η δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που τώρα είναι νεκρό γράμμα για την Βενεζουάλα με τις δολοφονίες που γίνονται, με τις παραβιάσεις και με τα ψέματα που ακούμε και τις απάτες. Ο Νίκολας ε, Μαδούρο εξεγελάει τους διεθνείς οργανισμούς μιλάει για κυριαρχία, μη παρέμβαση και εξού και δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Το 2013 όμως ε, υπήρξαν, υπήρξε δήλωση για 8.000 και δολοφονίες στο Κονγκό και έκανε κάτι ο Τώρα οι δολοφονίες αυξάνονται στη Βενεζουέλα. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν και εκεί για να διασφαλιστεί και εκεί η ειρήνη. Δεν μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα των διεθνών οργανισμών. Εμείς δεν θέλουμε να ζητιανέψουμε, δεν είναι κάτι τυπικό και κενά λόγια που λέμε. Όχι, θέλουμε η χώρα να βρεθεί και πάλι στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και χρειάζεται εξυγχρονισμός. Το Κοινοβούλιο δεν λέμε ότι θέλουμε να αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω από τα δικαιώματα του κράτους, θέλουμε όμως μηχανισμούς οι οποίοι να διευκολύνουν την εξίσωση που θα οδηγήσει στην κανονικότητα και όχι στις δολοφονίες και στη φτώχεια. Να υπάρξει και πάλι εξοπιστία στους θεσμούς και να αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι αδιαφορία. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να δημιουργούνται οι κατάλληλοι μηχανισμοί που θα καταπολεμήσουν τη βαρβαρότητα στη Βενεζουέλα. Και αν τα καταφέρουμε, θα είμαστε ευγνώμονες σε εσάς. Αν κάνετε και εσείς το χρέος σας. Πάντα θα σας ευγνωμονούμε για τη δράση σας που θα δώσει και πάλι ελπίδες στο λαό μας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, Ρώσο. Ε, Ευχαριστώ κι εγώ. Α, συγγνώμη, λάθος, λάθος. Ξέχασα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πω, πω, τι αγένεια από μένα. Είναι η πρώτη μέρα μετά τι διακοπές, βλέπετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα όσα έχω να πω, πιστεύω, θα καλύψουν ε, το σύνολο των ετοιμάτων θα επιθυμούσα επίσης να δώσω το λόγο κάποια στιγμή στον συναδελφό μου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το πολιτικό κομμάτι, για τα, δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παγίωση τη Δημοκρατία. Τα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικά φυσικά. Η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται εδώ και ένα χρόνο, όπως ε, είπαν και οι αναφέροντες. Πρόκειται για μια δραματική κατάσταση, την οποία γνωρίζουμε όλοι. Στη Βενεζουέλα μεταφράζεται σε μαζική μετανάστευση. Δραματική κατάσταση λοιπόν όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι κάνει η Κομισιόν, που είναι και ο στόχος της παρέμβασης μου εδώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε οπωσδήποτε ότι δεν υπάρχει πλέον δημιουργή συνεργασία με τη Βενεζουέλα. ως ε, χώρα μεσαίων εισοδημάτων. Το στρατηγικό έγγραφο λοιπόν ε, στο οποίο έγινε αναφορά είναι ένα έγγραφο αναφοράς από ανήκει όμως στο παρελθόν. Δεν ε, εφαρμόζεται πλέον, έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του, έχει τερματιστεί η εφαρμογή του, παρότι το περιεχόμενό του εξακολουθεί να ισχύει. Εξακολουθεί να αφορά πραγματικά γεγονότα. Τι κάνουμε τώρα, αφού δεν υπάρχει διμερή συνεργασία, συνεργαζόμαστε ουσιαστικά με αυτό που ονομάζουμε θεματικά προγράμματα που αφορούν τα, δικαιώματα των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και επίσης δράσεις ε, επισητιστικής ασφάλειας. Για να σας δώσω μια εικόνα, αυτή τη στιγμή ε, σε σχέση με τη Βενεζουέλα τρέχουν 15 ε, περίπου ε, συμβάσεις ύψου 8 εκατομμυρίων ευρώ τα 11 μαζί σε συνεργασία με τοπικέ ΜΚΟ. Σε θέματα λοιπόν υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουμε ουσιαστικά τους οργανισμούς υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ανθρώπου που μάχονται καθημερινά για τα, δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα υποστηρίζουμε και το ρόλο των νέων και των γυναικών μια διάσταση του φίλου δηλαδή. Για την κοινωνία των πολιτών, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Υποστηρίζουμε την παγίωση της κοινωνίας των πολιτών. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις δηλαδή, ουσιαστικά σε τομείς ε, που αφορούν τη διάσταση του φύλου, ε, την εξάλληψη των κοινωνικών αποκλεισμών, αλλά και την παροχή των βασικών υπηρεσιών. Όπως σημείωσαν οι αναφέροντες, υπάρχει ένα βασικότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την πρόσβαση της υπηρεσίας υγείας. Όπως επίσης και πρόβλημα διατροφικό. Επίσης έχουμε και κάποιες άλλες δράσεις υπέρ της ε, επιστημιστικής ασφάλειας που εκτελούνται σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Πέραν αυτού, επειδή η κατάσταση επιδεινώθηκε εδώ και περίπου δύο χρόνια, από πέρυσι ξεκινήσαμε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, όσο παράδοξο και να ακούγεται, σε μια χώρα όπως η Βενεζουέλα. Ανθρωπιστικές λοιπόν δράσεις ε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Βενεζουέλας. Υποστηρίζουμε διάφορες, ε, τις διάφορες μεταναστευτικές ροές. Ε, αυτή τη στιγμή μελετάμε τα επόμενα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 τα οποία προετοιμάζονται. Κάποια από αυτά θα υπογραφούν σύντομα κυρίως με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς. Αξίας περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ σε όλους αυτούς τους τομείς. Πριν κλείσω, να πω ότι έχουμε και κάποιες δράσεις περιφερειακών προγραμμάτων με τη Βενεζουέλα, αλλά η Βενεζουέλα ε, αδρανεί μάλλον στον τομέα αυτόν. Ο μόνο τομέα στον οποίο συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με αυτή τη χώρα είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τελείωσε ο χρόνο μου. Αυτό ήταν το BIP. Τώρα πριν ε, κλείσω να επαναλάβω ότι οι προσπάθειες που γίνονται εντός της Βενεζουέλας είναι εξαιρετικά δύσκολες. Αφενός διότι χρειαζόμαστε την άδεια ή τη σιωπηρή εξουσιοδότηση των αρχών για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Από την άλλη, δεδομένη τη οικονομική κατάσταση, είναι εξαιρετικά δύσκολη να διαχειριστούμε τον υπερβολικό πληθωρισμό, τον υπερπληθωρισμό. Ευχαριστώ. Τελείωσα. Αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε το λόγο στον συναδελφό μου. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο Κούτσεν Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν σχεδόν το όνομά μου. Ακούσατε εισαγωγικά τι προσπαθούμε να κάνουμε σε θέματα συνεργασία. Σήμερα η προσοχή εστιάζεται στη μεταναστευτική προσφυγική κρίση που βλέπετε σε όλη την περιοχή τη Νότια Αμερική, αλλά και στην Καραϊβική. Πολλοί μετανάστε έχουν φτάσει μέχρι και την Ισπανία και τι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν εμφανίστηκε σήμερα το πρόβλημα, ούτε πριν δύο χρόνια. Είχε ήδη ξεκινήσει, όπω αναφέρει ένα από του αναφέροντε, ε, εδώ και πολλά χρόνια. Πράγματι, αν διαβάσετε το έγγραφο 2017-2013, εκεί θα δείτε κάποιε από τι αδυναμίε του δημοκρατικού συστήματο που εντοπίστηκαν ήδη τότε πριν από 10 χρόνια στη Βενεζουέλα. Η κατάσταση πρώτα απ' όλα συνιστά πολιτική κρίση. Μια κυβέρνηση ε, ουσιαστικά καταχράστηκε της δημοκρατίας ε, προσπαθώντας να διατηρήσει την εξουσία και χρησιμοποίησε τον πολιτικό χώρο μόνο για τον εαυτό του χωρίς να αφήνει κανέναν άλλο στη χώρα. Γι' αυτό φεύγουν οι άνθρωποι, αλλά και λόγω της απουσίας φαρμάκων και τροφίμων, λόγω της οικονομικής πολιτικής ε, δεν υπάρχει πια τίποτα στη χώρα, γι' αυτό φεύγει ο κόσμος. Και ένας τρίτος λόγος που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η υψηλή βία και ατιμορρησία στη χώρα. Έχουμε ε, επίπεδα εκτιμόμενα, επειδή δεν έχουμε επίσημα στοιχεία, 30.000 δολοφονίες ετησίως το χρόνο ετησίω στη χώρα και κανεί δεν τιμωρείται, ούτε καν κατηγορείται, ούτε καν παρακολουθείται, ανακρίνεται για αυτά τα γεγονότα. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει διάφορε δηλώσει με κλήσει για την αποκατάσταση τη δημοκρατία, τη ε, κυβέρνησης, ε, μια σωστή κυβέρνηση για ένα σύνταγμα, για την απελευθέρωση, αποφυλάξη των ε, πολιτικών κρατουμένων και για την, να επιτραπεί ανθρωπιστική δράση σήμερα για τον τοπικό πληθυσμό και για όσους φεύγουν από τη χώρα. Εδώ και χρόνια ξεκινήσαμε με κάποια πρώτα σχόλια για την κατάσταση από τις καταστολές ε, των διαδηλώσεων του 2014 όταν ανέλαβε την εξουσία ο κ. Μαντούρο αλλά και τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλές δηλώσεις από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου επαναλαμβάνουμε διαρκώς τα ίδια και στα Ηνωμένα Έθνη στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των ΟΗΕ και εκεί έχει αναφερθεί πολλές φορές η κατάσταση στη Βενεζουέλα ε, με την υποστήριξη των χωρών της περιοχής. Θα συνεχίσουμε. Πριν από ένα χρόνο είχαμε κυρώσει για διαφορούς αξιωματούχους που θεωρούμε ιδιαίτερα υπεύθυνου για την πολιτική κατάσταση σε θέματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών του κράτους. Ήδη από πέρυσι επίσης έχουμε περίπου 18 άτομα σε αυτό το κατάλογο και έχουμε ε, ξεκινήσει και ένα εμπάργκο όπλων και για όλα τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή διαδηλωτών της αντιπολίτευσης. Διαρκώς λοιπόν παρακολουθούμε, μελετάμε, βρισκόμαστε σε διάλογο με τις ΜΚΟ, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και με εκπροσώπους της κυβέρνησης έχουμε διάλογο. Πάντα ελπίζουμε ότι κάποια μέρα θα ανοίξει ένα παράθυρο επικοδομητικού διαλόγου είναι πολύ περιορισμένες οι ελπίδε μα μετά από τις ε, πολύ κακέ εμπειρίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πάβουμε να διατηρούμε αυτή την πρόθεση να γίνει διάλογος. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε, να εφαρμόζουμε τις κυρώσει, μπορεί να εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων εάν καταστεί απαραίτητο και θα δούμε πώς μπορούμε να παρέχουμε περισσότερη ανθρωπιστική υποστήριξη στον πληθυσμό τόσο εντό τη χώρα εφόσον έχουμε πρόσβαση και για όσους διαφεύγουν από τη χώρα αυτή τη στιγμή στην Κολομβία, στο Περού, στην Χιλή, στην Αργεντινή και στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες. Η προσοχή μας λοιπόν εστιάζεται στην οικονομική βοήθεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κυβέρνηση αλλά ελπίζουμε ότι αυτή τη στιγμή με την υποστήριξη που παρέχουμε θα μπορέσουμε να ασκήσουμε κάποια πίσω ώστε να βρεθεί κάποια στιγμή κάποια λύση για τους ανθρώπους, για το λαό της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση των πραγμάτων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Και να σας ενημερώσω ότι ε, τούτη την ε, Πέμπτη η Επιτροπή Ντρουά θα έχει σχετική ακρόαση. Ρώσα, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους αναφέροντες. Εκείνοι μας παρουσίασαν στο πρώτο πρόσωπο πώς βλέπουν αυτή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, κράτους δικαίου και μια επιδείνωση όχι μόνο πολιτική αλλά και οικονομική και κοινωνική και ανθρωπιστική στη Βενεζουέλα. Οι Ισπανοί Έχουμε ιδιαίτερους ε, δεσμούς με τη Βενεζουέλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Οπότε είναι καλό που ήρθατε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήπειρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έρχονται από ολόκληρο τον κόσμο. Ακριβώς γι' αυτό και εμείς αυτό θέλουμε παντού στον κόσμο να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ειρήνη. Εξού και πριν από λίγα χρόνια βραβευθήκαμε με το βραβείο για την ειρήνη. Και ε, τώρα πρέπει να το κάνουμε πράξη αυτό. Πολλά ψηφίσματα έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το τελευταίο τον Ιούλιο που μας πέρασε, όπου εκεί αναφέρεται ότι υπάρχει ατιμορρησία στις περιπτώσεις βίας, ότι λείπουν τα πάντα φάρμακα, ότι δείκτες φτώχειας έχουν ανέβει φοβερά, τιμωρησία μετά από εγκλήματα, ότι ο λαός είναι πάρα πολύ ευάλωτος, ο κόσμος και μάλιστα ότι έχουν επανεμφανιστεί ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί, όπως είναι η λύσα, η μαλάρια κλπ. Υπάρχει και βέβαια μια τεράστια πολιτική κρίση. Συνεπώς, όπως πολύ σωστά είπε και η Πρόεδρος, το Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο. Έχουμε εργαστεί με τον συνάδελφο Αγγιλάρ στην Επιτροπή για τις Ελευθερίες του Πολίτη με τον κύριο Αγουστίν Μέρα, όλες οι πολιτικές ομάδες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως, οι αναφορές σας ακριβώς θα οδηγήσουν σε αυτή την κραυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να πιέσει πρότασή μου είναι να στείλουμε επιστολή στην είπα το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Μογκερίνη, για να μεταφέρουμε την ανησυχία και της δικιάς μας Επιτροπής, Επιτροπής Αναφορών, να στείλουμε επίσης επιστολή στην συνέλευση της Eurolat, προκειμένου και σε αυτούς να εκφράσουμε την ανησυχία της Επιτροπής μας και να στείλουμε επιστολή επίσης και στην Επιτροπή ε, ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκφράζοντας και εκεί την ανησυχία μας. Και βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλουμε επιστολή. Με αυτόν τον τρόπο θα μεταφέραμε ε, τους φόβους μας, τις ανησυχίες μας και την εκκλησία μας σε όλα αυτά τα θεσμικά όργανα. Και βέβαια θα ζητήσουμε και περισσότερες κυρώσεις γιατί μεταξύ άλλων εμποδίζεται και η ανθρωπιστική βοήθεια. Να μην υπάρχουν πια τέτοια εμπόδια στην Βενεζουέλα, ώστε τουλάχιστον ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να δοθεί και εκεί και στις γύρω χώρες. Καλώς ήρθατε, εν πάση περιπτώσει, στηρίζουμε τόσα είπατε. Και αυτή είναι η λύση που προτείνω αυτές τις δράσεις για να μπορέσουμε και να πιέσουμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Ευχαριστώ. Και εγώ χαιρετίζω με πολύ αγάπη τους αναφέροντες. Θα είμαι σύντομος γιατί χρειάζεται να επεκταθεί κανείς πολύ για να εκφράσει τη στήριξή του στις αναφορές αυτές που μας ήρθαν από πολίτες που ρητά λένε ότι είναι υπήκοοι και της Βενεζουέλας και της Ισπανίας, συνεπώς Ευρωπαίοι υπήκοοι. Στο άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, του Ισπανικού Συντάγματος, ε, αναφέρεται ότι υπάρχει διπλή υπηκότητα ε, για ανθρώπους ε, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, οι χώρες τους δηλαδή, με την Ισπανία, η Βενεζουέλα για παράδειγμα. Αυτό ισχύει και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτε και αυτό που μα φέρουν εδώ σήμερα είναι ένα σαφέ μήνυμα. Ζητούν τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου αυτό να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει, ε, να βρεθεί μια διέξοδος ε, για ειρηνική συνύπαρξη. Το λένε, το φωνάζουν, το κραυγάζουν. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για τη Βενεζουέλα εδώ στο σώμα και έχουμε εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα και σε αυτή τη θητεία που ολοκληρώνεται το Μάιο του 2019. Και μάλιστα το τελευταίο μας ψήφισμα ήταν στην τελευταία Ολομέλεια τον Ιούλιο του 2018. Δυστυχώς το ψήφισμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα είναι το τελευταίο, φοβάμαι, της θητείας αυτής, γιατί δεν φαίνεται να βελτιώνεται η κατάσταση εκεί. Οπότε, πέρα από την έγκριση των ψηφισμάτων μας που ζητούν διάλογο, περισσότερες προσπάθειες για μια δημοκρατική μετάβαση και ειρηνική στη Βενεζουέλα που να επιτρέψει στη χώρα να ξεπεράσει τα προβλήματά της και την κοινωνική ρήξη, τη βία, την ανασφάλεια, την προσωπική και τη συλλογική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυστυχώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω μα είπε και η ίδια η Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στη Βενεζουέλα, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ασκήσει διπλωματία. Και αυτό μέσω αυτού που λέμε soft power, ασύπιας δύναμη έτσι ευγενικά και διπλωματικά. Χρειάζεται όμως μεγάλη αποφασιστικότητα και άσκηση όλων των δυνατοτήτων μας προκειμένου οι κάτοικοι της Βενεζουέλας και πίκο της Βενεζουέλας που ζητάνε βοήθεια, καταφύγιο, ελπίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να έχουν και τις διπλωματικές μας προσπάθειες και τη συνεργασία μας για να ασκηθεί ε, πολιτική πίεση. Να ξέρουν ότι έχουν τη στήριξή μας ώστε να μπορέσει η Βενεζουέλα να βρει και πάλι την ειρήνη και την ειρηνική συμβίωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πισέρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες που ήρθαν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω εδώ την Πατρίθια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλε. Εμείς ε, γνωριστήκαμε στη Μαδρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ήρθε μετά από πολλά χιλιόμετρα που έκανε για να συγκεντρώσει τις χιλιάδες υπογραφές των Ευρωπαίων και να μας φέρει την αναφορά αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Μαδρίτη. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Πάντω, θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο τη υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης για τόσα μας είπε και για τις προσπαθίες τους. Ε, πράγματι, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γιατί αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα σήμερα, όπως και αν το ορίσει κανείς, δεν αποτελεί καρπό ε, φυσικής καταστροφής. Όχι. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πρόκειται μόνο για εκατομμύρια ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη χώρα, φεύγουν, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή, στη Βενεζουέλα συστηματικά και μεγάλη, με μεγάλη πολιτική ένταση χρησιμοποιείται η πείνα ώστε να πιεστεί ο κόσμος και να μπορέσει η κυβέρνηση να κρατηθεί στην εξουσία. Αυτή είναι αλήθεια και αυτό είναι που είναι ντροπή. Όταν μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση, βεβαίω και υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Και εδώ αρχίζουμε να δρούμε, γιατί έχουμε τρόπο να δράσουμε, στα σύνορα της Βενεζουέλας, γιατί μέσα στη χώρα δεν μπορούμε να πάμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πίσω πόρτα, από το παραθυράκι, αλλά υπάρχει από το καθεστώς του Μαδούρο συστηματική άρνηση. Και αυτό είναι ένας από τους παράγοντες, ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα τα 7 κατά της ανθρωπότητας που αναφέρει η έκθεση τριών εμπειρογνωμόνων υψηλού κύρους που συνέταξαν εκ μέρους ε, των Αμερικανικών ε, κρατών, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών. Ελπίζω από βάθους καρδίας οι ευρωπαϊκές χώρες να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στα δικαστήρια, στο πυρικό δικαστήριο, γιατί είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας να χρησιμοποιεί ένα καθεστώς την πείνα του κόσμου για να κρατηθεί στην εξουσία. Είναι έγκλημα. Δεν ξέρω αν κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Η πολιτική θέση και βούληση υπάρχει, οι κυρώσεις υπάρχουν. Ας ελπίσουμε ότι θα ενισχυθούν οι κυρώσεις, θα τεθούν σε εφαρμογή πλήρως. Και κατά τα άλλα αυτή η εξαιρετική ανθρωπιστική βοήθεια που δόθηκε τα 5 εκατομμύρια για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη χώρα και που βρίσκονται σε πάρα πολύ σοβαρή ε, κατάσταση υγιεινής πρώτα απ' όλα, βοηθούνται. Αλλά επιπλέον οι χώρες μέλη έχουμε την υποχρέωση κατά τη γνώμη μου, δεδομένου ότι έχουμε υπογράψει τη Ρώμη, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να ζητήσουμε από το ποινικό δικαστήριο να ξεκινήσει έρευνα, γιατί αυτά είναι εγκλήματα τα οποία δεν παραγράφονται. Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε πολιτικά, εντάξει, και η Κομισιόν ε, τα λέει και τα κάνει και έχει τις δυνατότητες να κάνει αυτά που κάνει. Γιατί σας λέω υπάρχουν χιλιάδες Βενεζουελάνοι που βρίσκονται στην Ευρώπη και είναι και Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα είναι κάτι που έχει να κάνει και με τους δικούς μας πολίτες, έτσι, τους Ευρωπαίους. Αλλά επιπλέον Οι δράσεις των χωρών μελών που πρέπει να κάνουν πρέπει να, που τις, πρέπει να τις κάνουν όλοι και Ισπανία ακόμα περισσότερο, πρέπει να φροντίσουν για δικαιοσύνη, ανθρωπιστική βοήθεια, δικαιοσύνη και ξανά δημοκρατικό σύστημα στην Βενεζουέλα. Αυτά είναι τα πεδία δράσης μας. Οι αναφορές αυτές που θα πάνε και στον κύριο Λαμπρινίδη και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κλπ. για να αποφανθούν όλοι αυτοί. Αλλά επιπλέον να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να έχουμε την απάντηση του κύριου Λαμπρινίδη. Γιατί αυτά που γίνονται στη Βενεζουέλα θα επιδεινωθούν. Οπότε είναι υποχρέωσή μας να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα διαθέτουμε και ό,τι παράθυρα μπορούμε να ανοίξουμε ώστε να συνεισφέρουμε γιατί είναι χρέος μας να το κάνουμε. Ευχαριστούμε, Τερεκάμπρας. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες που ήρθαν με κάθε σεβασμό. Είναι αλήθεια ότι μας φέρνουν τον πόνο τους και την απελπισία τους σε ένα μεγάλο βαθμό. Όμως κάποια στιγμή ανησύχησα λίγο κυρίως από αυτά που άκουσα από τη δεύτερη παρέμβαση, που από αυτά φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Και ότι σήμερα ήρθαν να μας πείσουν και σήμερα θα αρχίσουμε εφόσον μας πείσουν. Και αν δεν μας πείσουν, μεγάλη καταστροφή. Αυτό ήταν το πνεύμα. Με τους συναδέρφους μπορεί να έχουμε πολιτικές διαφορές, ιδεολογικές κτλ. Τους δεν θα μπω μέσα σε αυτό. Όλοι μιλήσανε για την ανθρωπιστική καταστροφή. Ανθρωπιστική καταστροφή, συνεπώ όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και το υπενθύμησαν και οι συνάδελφοι και η Κομισιόν ότι ψηφίσματα πολλά έχουμε εγκρίνει, ότι έχουμε βραβεύσει και την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, αυτούς που αγωνίζονται δηλαδή για την αλλαγή κλπ. Οπότε η δράση μας δεν ε, μετράει εφόσον μας λέτε ότι δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άρα ούτε και εμείς μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κι όμως δημιουργείται αίσθηση, υπάρχει ηθική στήριξη. Όπως υπενθύμισε και ο συνάδελφος Λόπες Αγγελάρ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει εξουσίες πάνω σε αυτό το θέμα. Και η δικιά μας Επιτροπή δεν έχει ούτε εκτελεστικές αρμοδιότητες, ούτε μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Μπορούμε να καταδικάσουμε, να καταγγείλουμε και το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να λυθεί η υπόθεση, που θα λυθεί όμως με τρόπο που πολύ μπορεί λίγο πολύ να φανταζόμαστε, αλλά που κανένας δεν ξέρει ακριβώς πώς για να υπάρχει ειρήνη κλπ. Πρέπει να είμαστε όμως ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Εσείς προσπαθείτε, όπως και εγώ θα προσπαθούσα παντού στον κόσμο, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε την εξουσία, την αρμοδιότητα, ούτε τις δυνατότητες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούμε τις εκκλήσεις σας και την κραυγή που μας φέρνετε. Η Ρώσα. Δεν συμφωνώ ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να κάνει πολλά, μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Και θέλω να το πω και το είχα πει στον κύριο Τερεσκάβρα τότε που είχαμε την ε, συζήτηση για τα παιδιά που έχουν απαχθεί. Κι όμως κάνουμε την αλλαγή. Είναι ένα όργανο που μπορεί να πιέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας και μπορεί Λοιπόν, την προηγούμενη φορά εσύ με έπεισε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Τώρα ελπίζω να σε πείσω εγώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Εσύ με έπεισε τότε που ασχοληθήκαμε με τα παχθέντα παιδιά χωρίς να έχουμε την αρμοδιότητα. Όταν ασχοληθήκαμε με το ατύχημα, χωρίς να έχουμε αρμοδιότητα. Χιλιάδες φορές χωρίς να έχουμε αρμοδιότητες ασχοληθήκαμε και ο συνάδελφος με έπεισε. Τώρα λοιπόν εγώ θέλω να τον πείσω ότι μπορεί να μην έχουμε αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να βρωτοφωνάξουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα και ότι πρέπει να βρεθεί ειρήνη. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, δεν θέλω να ξεκινήσουμε διάλογο για το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα θέλω να ξεκαθαρίσω και πρέπει να διορθώσω και τους δυο σας. ότι έχει, ό,τι και να έχει γίνει στην Ισπανία, είτε αφορά τα βρέφη είτε διποτε έχει γίνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Βενεζουέλα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακούσαμε ε, από την ΕΕ τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμή. Επίση, οι αναφορέ αυτέ έχουν διαβιβαστεί από την Επιτροπή Αναφορών στην ΤΡΟΑ, που είναι η υποεπιτροπή τη ΑΦΕΤ που θα οργανώσει ήδη τώρα την 5η 6 Σεπτεμβρίου ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα και την Κούβα. Συνεχίζονται οι εργασίες ε, στην Επιτροπή αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα. Η δική μας Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει πολλά, αλλά παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος. Θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο στους αναφέροντες. Πολύ σύντομα, δύο λεπτά ο καθένας. Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις και συμφωνώ με τον κύριο Τέρα Κάμπρες. Ναι, μία αναφορά μπορεί να μην μπορεί να κάνει πολλά πράγματα πέρα από μια κραυγή, αλλά πολλές κραυγές μαζί κάνουν μια αλλαγή. Και θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουν τα πράγματα επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάτι. Δεν είναι αυτό που λέμε. Αλλά πρέπει να γίνει γνωστό. Ο κόσμος είναι πολύ πιο μικρό σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Ό,τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, επηρεάζει αυτά που συμβαίνουν εδώ. Ό,τι γίνεται στη Συρία, επηρεάζει την κατάσταση εδώ. Ό,τι γίνεται στην Καμπόν, επηρεάζει την κατάσταση εδώ. Ε, και με εμά το ίδιο ισχύει. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσει η κατάστροφη όπως έγινε στη Ρουάντα, στο Κονγκό, να έχουμε 3-5 εκατομμύρια και μετά να λέμε κάτι έπρεπε να είχαμε κάνει. Δεν λέω ότι έχω εγώ την απάντηση. Δεν έχω την απάντηση τι μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την πίεση που προωθείτε τις αναφορές μας αυτούς που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Πρώτα απ' όλα την ε, κυρία Μπεθέρα. Γιατί πραγματικά είναι ηρωίδα για τους Βενεζουελάνους πέρα από οποιαδήποτε ιδεολογία, τις βγάζουμε το καπέλο. Πιστεύω, ή είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, με κάθε σεβασμό. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό κόμμα. Είμαι ανεξάρτητη και είμαι μητέρα ε, από τη Βενεζουέλα, ε, δικηγόρος και ακούω τις φωνές όλων που φωνάζουν «Βοηθήστε». Χιλιάδες έχουν υπογράψει πάνω από 67.000 υπογραφές που ζητούν μάλιστα και ανθρωπιστική διαδρομή για να πηγαίνει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πράγματι, έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα πέρυσι μέχρι να φτάσει η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι περιμένουν κάποια βοήθεια. Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάθε σεβασμό να προθίσει την αναφορά μας στο ποινικό δικαστήριο, στην εισαγγελία, στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, το Γενικό Γραμματέα, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν περιμένουμε μόνο όμως θεσμική βοήθεια. Ό,τι μπορούν να κάνουν οι θεσμοί, αλλά και εμείς οι πολίτες βοηθούμε τη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Άννα, πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση για να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην γίνεται γενοκτονία όπως γίνεται τώρα στη Βενεζουέλα, πάνω από 27.600 δολοφονίες πέρυσι και πρόπερση Πού να ζητήσει κανεί αυτή την μεταρρύθμιση, αν δεν τη ζητήσει εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν πρέπει να υπάρχει κάποια μεταρρύθμιση του νόμου, ένα γίνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας διαβεβαιώ, κυρία Καρέρα Ρόχα, ότι έχει ακουστεί η έκκλησή σας και έχει απαντηθεί από την Επίτροπή μας, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Ακούσατε τα ψηφίσματα που ήδη έχουν εγκριθεί και με την πλήρη υποστήριξη του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναλάβει περαιτέρω δράση. Επίσης, η Επιτροπή μας έχει διαβιβάσει τις αναφορές στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Και επαναλαμβάνω τρίτη φορά ότι σε δύο μέρες από τώρα θα έχουμε και τη σχετική ακρόαση. Αυτό έχει κάνει η Επιτροπή μας και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Σας ακούσαμε. Ναι, πρόκειται για εφιαλτική κατάσταση. Η ανθρωπιστική μας υποστήριξη και η κατανόησή μας ε, είναι δική σας. Τώρα εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα επανέλθει στο θέμα αυτό. Ετούτη τη στιγμή, μετά από όλα ήδη έχουν γίνει, μπορούμε να στείλουμε επιστολή στην Φρεντερίκα Μογκερίνη, όπου να συνοψίζουμε αυτά που είπατε και την συζήτηση στην Επιτροπή μας και να κλείσουμε την αναφορά. δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ όμως πολύ ευχαρίστω σας συντάξω αυτήν την επιστολή προσωπικά. Συμφωνεί η Επιτροπή να προχωρήσουμε με τον τρόπο αυτό. Εξαιρετικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε μέχρι εδώ. Από τη Βενεζουέλα ήρθατε αν δεν κάνω λάθος. Και εσείς. Όχι, εγώ μένω στο Ρότερνταμ. Σας ευχαριστώ όλους. Όσοι ήρθατε εδώ, όσοι ταξιδέψατε από πιο κοντά ή από πιο μακριά και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον. Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση δείχνοντας κάθε κατανόηση και σε προσωπικό επίπεδο. Σας εύχομαι ασφαλή επιστροφή. Ευχαριστώ την ΕΙΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα τη σημερινή ημερησίας διάταξης που είναι το σημείο 10 έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2017. Η συγγήτρια είναι η κυρία Εύη. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 6 του μήνα, την 5η στις 3. Και θα ψηφίσουμε τον Νοέμβριο. Τούτων λεχθέντων, ας ακούσουμε την Ελεονόρα, παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά την Ευρωπαϊκή Δημοσιολαβήτρια για τη δουλειά της. Το αναφέρω και στην αρχή της έκθεσης. Στην έκθεση αυτή ήθελα να δώσω ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες σοβαρές επικρίσεις ε, που υπήρξαν αντικείμενο των ερευνών για τη διαμεσολαβήτρια η μη διαφάνεια των, ε, της λήψης αποφάσεων, τα ηθικά προβλήματα που περιέλαβαν και εν ενεργεία επιτρόπους, τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον σημερινό πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ένα νομικό πλαίσιο που έχει κενά ε, δεν παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων ε, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας από τα λόμπι. Όλα αυτά υπονομεύουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και την λυπή ε, ε άδεια πρόσβασης στα έγγραφα από τους ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούν να ασκήσουν έτσι τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Έχω υπογραμμίσει επανειλημμένως στη στη Λαβήτρια ότι υπάρχουν επικρίσεις ε, και κάποιες επικοδομητικές συστάσεις για βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου. Ωστόσο, υποχρεωμένα να διαπιστώσω με δυσαρέσκεια και ανησυχία ότι οι απαντήσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι μη ικανοποιητικέ, ε, εξωφρενικές μερικές φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να πέφτει σε μια άβυσο αναξιοπιστίας και δυσπιστίας των πολιτών της, επειδή δεν αλλάζει η ηθική πολιτική και οικονομική στάση. Έχουμε την περίπτωση Μπαρόσου που στο τέλος της θητείας του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διορίστηκε μη εκτελεστικός πρόεδρος και σύμβουλος της ε, ε τράπεζας Goldman Sachs που ενεπλάκη στην ε, οικονομική κρίση του 2008 μεταξύ άλλων. Τότε ε, υπόθηκε ότι υπήρχε κακή διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόθεση αυτή. Η, η Επιτροπή Διοντολογίας εντός της Κομισιόν λόγω της μη ανεξαρτησία από το πολιτικό επίπεδο συμπέρανε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν παραβίαση νομικών υποχρεώσεων από τον Παρόσο και απλά έλαβε υπόψη μια δήλωση γραπτή του Μπαρόσο που δήλωνε ότι δεν τον είχε ε, πάρει η Goldman Sachs για lobbying. Αλλά το Σεπτέμβριο του 2017 ανακαλύφθηκε αντιθέτω ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Μπαρόσο και του σημερινού Αντιπρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κ. Κατάινεν, που καταγράφηκε ω επίσημη συνάντηση με την Goldman Sachs. Η φύση τη συνάντηση, όπω λέει η δημοσιολαβήτρια στην έρευνά τη, δεν είναι σαφή και δημιουργεί ανησυχίε για το ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαρόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει την πρώην ε, θέση του και τις επαφές του για να επηρεάσει τα πράγματα ή να δώσει πληροφορίες ή για να εκτελέσει ε, εργασίε lobbying για την Goldman Sachs. Μια άλλη προβληματική περίπτωση του 2017 είναι αυτή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, στην ομάδα των 30, μια, έναν ιδιωτικό οργανισμό που έχει εκπροσώπους τραπεζών που υφίστανται ε, επιτήρηση από την Κεντρική Τράπεζα. Η συγκήτρια ζήτησε από τον πρόεδρο της ε, Κεντρικής Τράπεζας να μην συμμετέχει σε αυτή την ομάδα, αλλά μέχρι σήμερα έχει αρνηθεί. Κατά την άποψή μας, ε, αυτό αμαυρώνει την εικόνα ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα έπρεπε να είναι και να φαίνεται ανεξάρτητη από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Όσον αφορά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατηρείται η μη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων. Δεν υπάρχει πρόσβαση για το κοινό σε αυτούς τους διαλόγους, δεν υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες του Συμβουλίου, δεν καταγράφονται οι θέσεις των κρατών μελών στα φάιλ και απορρίπτονται όλες οι αιτήσει πολιτών να δουν τα έγγραφα. Η Διαμεσολαβήτρια το 2017 κατήγγειλε καθαρά αυτές τις συμπεριφορές του Συμβουλίου ως κακοδιαχείριση. Το 2018 ακολούθησε η ειδική της έκθεση εστιασμένη στα ειδικά προβλήματα διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου. Το status quo έρχεται σε αντίθεση με τη νομική κατεύθυνση που έδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που επανέλαβε στην απόφαση της 22ης Μαρτίου του 2018 στην υπόθεση Καπιτάνη ότι οι αρχές διαφάνειας και δημοσιοποίησης είναι εγγενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να μην εφαρμόζονται πλήρω για λόγους ε, αποτελεσματικότητας όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Η έλλειψη πληροφόρησης για την νομοθετική διαδικασία δεν αποτελεί απλά παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά εντείνει και τη δυσπιστία τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται και λόγω της μη αναθεώρησης ε, του κανονισμού 1049 του 2001 που έχει σχέση με την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, ε, του οποίου οι διατάξεις έχουν ε, πλέον θεωρούνται απερχαιωμένες. Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Όσον αφορά τη διαφάνεια, για τη χρήση, με τη χρήση της φράσης full transparency που θα βρείτε πολλές φορές στο κείμενο θέλησα να τονίσω ότι πρέπει να μειωθεί η διακριτική ερμηνεία από τα θεσμικά όργανα που συστηματικά εξακολουθούν να απαγορεύουν στους πολίτες να δουν τι επιλογές έχουν γίνει στα θεσμικά όργανα και τι διαδικασίε έχουν ακολουθηθεί. Είναι απαράδεκτο να μην ακολουθείται ένα μητρό υποχρεωτικό ε, διαφάνειας ε, τόσο για τον τομέα τον ιδιωτικό όσο και για τα θεσμικά οργάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να παρακολουθούνται οι δραστηριότητες lobbying. Επίσης δεν είναι αποδεκτό το ότι Ακόμα είναι αδιαφανείς οι πληροφορίες όσον αφορά τις ε, περιστρεφόμενες πόρτες ώστε να γνωρίζουμε τα ονόματα των ε, υπαλλήλων που ξαφνικά φεύγουν από τα θεσμικά όργανα και βρίσκουν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Είναι απαράδεκτη η εφαρμογή τη ασχή τη μη αποκάλυψη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για πληροφορίε και έγγραφα που έχουν συλλεχθεί σε ε, περιπτώσει ελέγχων και ερευνών, ακόμη και σε περιπτώσει απάτη ή διαφθορά, όπω στο Dieselgate. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει απόλυτη καθαρότητα και ανεξαρτησία από τον ιδιωτικό τομέα κατά τη συλλογή και την αξιολόγηση των επιστημονικών στοιχείων που πρέπει να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όπως για παράδειγμα έγινε στην περίπτωση της έγκρισης για τη συνέχιση της χρήσης ε, της γλυφωσάτης αλλά και άλλων ε, ε, ουσιών γενετικά τροποποιημένων και φυτοφαρμάκων. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει μια στρατηγική έρευνα. Έχω ολοκληρώσει την παρουσίασή μου. Θα ήθελα να έχω τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων για να βελτιώσουμε το κείμενο αυτό και είμαι βέβαιη ότι θα το καταφέρουμε σε ένα πνεύμα συνεργασίας που ανέκαθεν διέκρινε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ πολύ, ο Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση που έχει συντάξει η συνάδελφος η κυρία Ήβη. Θα ήθελα να θέσω ορισμένα θέματα. Στα περισσότερα συμφωνούμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ρόλο που έχει επιλέξει και πολύ σωστά η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο ή με τις αποφάσεις της επηρεάζει την καθημερινή ζωή ε, των πολιτών αλλά βεβαίως και όλης της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως πρέπει να είναι ανοιχτή στον έλεγχο, να έχει διαφάνεια και αυτό αφορά όχι μόνο τη συμμετοχή του κυρίου Ντράγκη στη γνωστή ομάδα των 30, ε, αλλά βεβαίως και όλη τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το γεγονός ότι ο κύριος Ντράγκη επιμένει να παραμένει σε αυτή την ομάδα των 30 όπου συμμετέχουν και τράπεζες που βρίσκονται υποτίθεται κάτω από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι που δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στα θέματα ελέγχου. Δεύτερον, θεωρούμε σημαντική την παρέμβαση της Μεσολαβήτριας στην υπόθεση του κυρίου Μπαρόζο απεδείχθη ότι πλέον έκανε συνάντηση εκ μέρους της Goldman Sachs με τον κύριο Κατάινεν, ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε βεβαίως και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το τρίτο θέμα αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη διαφάνεια και να επισημάνω αυτό που έχω πει επανειλημμένα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι η συγκεκριμένη τράπεζα έδωσε 230 εκατομμύρια ευρώ δάνειο στη Fraport προκειμένου να συγκεντρώσει το ποσό που απαιτείται για την αγορά και τις επενδύσεις στα ελληνικά 14 αεροδρόμια. Η Fraport έπρεπε να καταβάλει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να για τα ελληνικά αεροδρόμια τα 14 έχει μαζέψει πάνω από 950 εκατομμύρια ευρώ από δάνεια και 230 εκατομμύρια ευρώ τη έδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για μένα δεν είναι σοβαρός επενδυτής η Fraport. Αυτό που ισχύει είναι ότι στηρίχθηκε πλέον από τις τράπεζες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το επόμενο θέμα που είναι ιδιαίτερα σοβαρό αφορά τη λειτουργία του Eurogroup διότι το Eurogroup είναι κράτο εν κράτη, παίρνει αποφάσει που επηρεάζουν καθημερινά την λειτουργία των πολιτών, έχει διαλύσει την οικονομία τη Ελλάδο, αλλά και του Νότου με τι αποφάσει που έλαβε. Έχουμε τον κύριο Ντάισεμπλουμ ο οποίο ομολόγησε ότι οι αποφάσει που πήραν στο Eurogroup για την Ελλάδα δεν βοήθησε του Έλληνε πολίτε, αλλά διέσωσε τι τράπεζε και του ξένου επενδυτέ. Δεν μπορεί να είναι στο απειρόβλητο το Eurogroup και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει συστηματικό έλεγχο και πολιτικός αλλά βεβαίω και τη κακοδιοίκηση, η οποία υπάρχει στο Eurogroup καθώς δεν υπάρχει διαφάνεια και η έλλειψη διαφάνειας σημαίνει κακοδιοίκηση. Κλασική περίπτωση εκδίδει τις αποφάσεις του μόνο στα αγγλικά όταν οι αποφάσει του αφορούν την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και δεν υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις στις γλώσσες των κρατών που αφορούν οι αποφάσεις του Eurogroup. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στον, τριμερή διάλογο δεν καταγράφονται οι θέσεις των κρατών μελών δηλαδή των κυβερνήσεων που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία και έτσι κανείς δεν ξέρει τι είπαν συγκεκριμένα κόμματα εξουσίας ε, σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο Συμβούλιο. Πολύ δε περισσότερο καθώς πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές που πρέπει να υπάρξει διαφάνεια. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουμε τι λέει ο καθένας και τι ψηφίζει. Το ίδιο πρέπει να ξέρουμε και να ισχύει και για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Για τα υπόλοιπα θέματα θα υποβάλουμε και εμείς ε, τροπολογίες ε, στην έκθεση της συναδέλφου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now, let's see. Ο Πίτερ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την εισηγητρία. Δεν ξέρω να ξεκινήσω από τα καλά ή τα κακά Θα ξεκινήσω από τα καλά. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τη διαμεσολαβήτρια όσον αφορά την διαφάνεια. Υπάρχει μια δυσαναλογία ε, όταν κοιτάμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και πώς λαμβάνονται εκεί οι αποφάσεις. Γνωρίζω ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε, αλλά συμφωνώ με τη διαμεσολαβήτρια. όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας θα πρέπει να δημοσιεύει κανείς τη θέση του και την αιτιολόγηση της ψήφου. Εγώ ως ε, Γερμανός πάντα δυσαρεστούμε όταν βλέπω να επικρίνονται οι Βρυξέλλες ε, αλλά στην Γερμανία να πρέπει να εξηγήσω ότι και τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στις ψηφοφορίες των Βρυξελών. Αλλά έχουμε και την άλλη πλευρά. Δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικά πολύ διαφάνεια που να εμποδίζει τη διεξαγωγή των εργασιών. Το διαδίκτυο είναι κατά 200% διαφανές, αλλά πάλι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Εγώ όλη μέρα μιλώ με λομπίστες, μιλώ με τους ενδιαφερομένους, συμπληρώνω το σχετικό έντυπο, αλλά θα πρέπει η διαφάνεια να εφαρμόζεται με τρόπο αποδεκτό. Θα πρέπει να βελτιώσουμε όχι τη στατιστική, αλλά την πραγματικότητα, διότι μερικές φορές έχουμε απλά καταπολέμηση της ε, έλλειψης διαφάνειας στο χαρτί, όχι όμως στην πραγματικότητα. Και όταν μιλώ με λομπίστες, ε, ότι ε, πολλά πράγματα δεν θα ήταν δυνατά διαφορετικά. Επόμενη παρατήρηση. Πιστεύουμε ότι στην έκθεση θα πρέπει να αναφερόμαστε στην διάκριση των αρμοδιοτήτων διαμεσολαβήτριας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέλος, στις τελευταίες εκθέσεις αναφέρεται πάντα η υπόθεση Μπαρόσο. Η έκθεση όμως είναι αιτήσια. Πώς είναι δυνατόν να ανακύπτει συνέχεια η, η ίδια περίπτωση. Ωραία, συνέβη αυτό, δεν ήταν ωραίο. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερους κανόνες. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχει λήξει η υπόθεση Βαρόσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα υποβάλουμε τροπολογίες. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κύριε Τσουφρίντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της ε, μεγαλόπνοη. Και έτσι θα είναι και οι προσπάθειες που θα ακολουθήσουν φιλόδοξες, ε, διότι είναι σημαντικό αυτό. Η μορφή της διαμεσολαβήτριας είναι σημαντική και η λειτουργία της επίσης. Πραγματικά σημαντικός πόρος, ειδικότερα όσον αφορά τις περιπτώσεις ε, και υποθέσεις ε, κακοδιαχείρισης. Δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω στους συναδέλφους μου. Με ένα κομμάτι από όλα αυτά συμφωνώ τα στοιχεία είναι αδιάσυστα όλα αυτά που βλέπουμε στην έκθεση της εισηγήτριας. Ελάχιστο περιθώριο ερμηνείας υπάρχει η παρανόηση. Πράγματι, τα σημαντικότερα ζητήματα ε, στα οποία επικεντρώθηκαν οι έρευνε τη Δεμεσολαβήτρια που αρχιοθετήθηκαν το 2017 ήταν η διαφάνεια, η πρόσβαση στα έγγραφα, ε, τρόπο παροχή τη υπηρεσία και οι διαδικασίε. Πολλά πράγματα εξακολουθούν να πρέπει να διορθωθούν και να επιληθούν. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό άφοβα να προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που αναφέρει η έκθεση και τα οποία συζητήθηκαν και σήμερα. Όλες αυτές τις υποθέσεις όπως για παράδειγμα των περιστρεφόμενων θυρών, την απροθυμία ε, του Συμβουλίου σε πολλέ περιπτώσει όπω είδαμε, κατάφορες περιπτώσεις. Θέλουμε το Συμβουλίο να βελτιώσει τη διαφάνεια των συνεδριάσεών του, να δημοσιεύει αν μη τι άλλο τα έγγραφα κλειδιά των τριμερών διαλόγων όπω ζήτησε και η Όχι όλα, είναι αδύνατον, αλλά αν μη τι άλλο σίγουρα τα σημαντικά, τα καθοριστικά. Επ' αυτού θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μας στην έρευνα και τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα του Συμβουλίου που θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όσον αφορά τι δικέ μου τροπολογίε και σε αυτή και σε άλλε περιπτώσει, όπω είπα, θα ήθελα τα αιτήματα να εμπνέονται από την πεποίθηση ότι ε, η καλύτερη γνώση των θέσεων των εθνικών κυβερνήσεων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα μειώσει την νοοτροπία του να κατηγορούμε διαρκώ τι Βρυξέλλε, τον blame Brussels. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό διότι σχετίζεται, αφορά τη σχέση των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλει στην παραπληροφόρηση που σήμερα χαρακτηρίζει τα πάντα που λέγονται γύρω από τα, Ευρω... από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής για τη Χρήση των Φυτοφαρμάκων και της Επιτροπής Γεωργίας και γι' αυτό υποστηρίζω θερμά την έκκληση προς τη Διαμεσολαβήτρια να κάνει ε, ό,τι μπορεί για να γίνει σύντομα έρευνα αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της Ένωσης διασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση και η εξέταση των επιστημονικών στοιχείων γίνεται διαφανώς και ανεξάρτητα, ειδικότερα όσον αφορά τη γλυφοσάτη, υλικό για το οποίο γίνονται πολλές συζητήσεις σε πολλές επιτροπές. Δυστυχώ δεν αρκεί ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μα. Έτσι κλείνω Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα πριν κλείσω να ευχηθώ καλή δουλειά και να συγχαρώ ε, εκ μέρους ε, των σοσιαλιστών την Έμιλιο Οράιλη για τις προσπάθειές της και για την επιμονή που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της και τη δουλειά της. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έχω μία ερώτηση κάπως ε, λεπτή. Δεν έχω αντιπρόεδρους εδώ όπως βλέπετε. Η Ευρωπή με έχει βοηθήσει γιατί εγώ πρέπει να προευρεθώ σε μια άλλη πολύ σημαντική συνάντηση. Θα ήθελα να με αντικαταστήσει κάποιος και τώρα κοιτάω τις ηλικίε σας συνάδελφοι για να ζητήσω από τον γυρεότερο. Κύριε Τερικάμπρας, εσείς είστε ο μεγαλύτερος σε ηλικία, αλλά μη με κοιτάτε έτσι, λέει ο κύριο Τερικάμπρα. Αλλά τώρα εδώ μπαίνει το λεπτό στοιχείο τη παρέμβασή μου. Είστε όμως εισηγητής του επόμενου σημείου. Θα ήθελα να σας καλέσω λοιπόν. Με άλλα λόγια λοιπόν ψάχνω τον δεύτερο γυρεότερο, ο οποίος είναι ο Πίτερ Γιάρ. Θα είχατε την καλοσύνη να έρθετε να με αντικαταστήσετε για ε, δύο επόμενα σημεία. Όχι, όχι, λέει η πρόεδρος. Ε, μια χαρά θα τα καταφέρετε. Μπορώ. και να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποστήριξή σας. Η Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Βρισκόμαστε στο τέλο ε, του σημείου αυτού τη ημερησίας διάταξη και γι' αυτό δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στην συνάδελφο Εύη για τι τελικέ της παρατηρήσει. Ε, δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή. Bene, ehm, Ωραία, ήταν πολύ σύντομη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνοψίσω λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Πολύ ευχαρίστω θα ακούσω τις παρατηρήσεις τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι σημαντικό για μένα είναι να εξετάσουμε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που έχει θίξει η διαμεσολαβήτρια και τα θέματα που ανέφερε ο συνάδελφος Μαριάς, ε, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurogroup. Αυτά δεν συμπεριλαμβάνονταν στην έκθεσή μου. Νομίζω όμως ότι γενικά υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την προσέγγιση μας ε, όσον αφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο. Επίσης, όσον αφορά την προσέγγισή μας στη διαφάνεια αυτή καθ' αυτή, Άκουσα ότι ο συνάδελφος Γιάρ έθιξε ένα θέμα σημαντικό. Η διαφάνεια θα πρέπει να είναι ο γενικός κανόνας και μπορούν κατόπιν να υπάρξουν εξαιρέσει στον κανόνα αυτό όταν υπάρχει ανάγκη προστασία συγκεκριμένων δεδομένων. Σήμερα όμως, αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ακριβώς το, αντίθετο. Θα πρέπει λοιπόν η διαφάνεια να είναι ο κανόνας και να υπάρξουν εξαιρέσει και όχι το αντίστροφο. Αυτό λοιπόν λέω στο σχέδιο εκθεσή μου. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και περιμένω με χαρά να δω τις ε, τροπολογίε του και προσλέπω στη συνέχιση των εργασιών ε, στο πνεύμα συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Υποθέτω ότι και οι συνάδελφοι θα δράξουν την ευκαιρία να υποβάλουν τροπολογίε. Ε, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το σχέδιο γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή του χάρτη των θεμελιωδών ε, ε, δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θεσμικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 7η Σεπτεμβρίου στι 3 ώρα το απόγευμα. Πρώτα όμω δίνω το λόγο στον εισηγητή Γιώσεπ Μαρία Τέρι Κάμπρας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. That. Well, well. Uh, uh, Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά κατηγορείται για πολυπλοκότητα, για διαφορία από τους πολίτες της. Το γεγονός ότι ο χάρτης ισχύει μόνο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αυτά εφαρμόζουν ε, δυνάμει του άρθρου 51 την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θεωρείται ανεπαρκές και μη ικανοποιητικό για πολλούς πολίτες. Η κατάσταση δημιουργεί περισσότερη αποξένωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να βελτιώσουν το πεδίο εφαρμογή του χάρτη. συνολικά ουσιαστικά διαφωνούμε με την Κομισιόν όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 51.1 που αξιολογεί διάφορες ε, αναφορές ε, που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο. Το σχέδιο πρότασης απευθύνει έκκληση και στην Κομισιόν ώστε να εισάγει μία εκτίμηση αντικτύπου των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις νέες ε, σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Δεύτερον, να ε, συμβουλεύεται τακτικά ε, την υπηρεσία θεμελιδών δικαιωμάτων όταν τίθεται θέμα θεμελιδών δικαιωμάτων. Τρίτον, να υποστηρίζει μια υποχρεωτική αξιολόγηση και αναθεώρηση των κρατών μελών όσον αφορά τη τήρηση των διατάξεων του χάρτη, κυρίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πριν κλείσω, σας καλώ να υποβάλλετε τροπολογίες για να συμπληρώσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Τα υποβάλλω και εγώ ενδεχομένως, ώστε να συμπληρωθούν ορισμένε πτυχέ δεδομένου του περιορισμένου χώρου που έχουμε για τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαριάς θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να συγχαρώ τον συνάδελφο, τον κύριο Τερικάμπρας, για την έκθεσή του. Συμφωνώ στα περισσότερα σημεία. Θα προσθέσουμε και εμείς ορισμένες τροπολογίες, αλλά θέλω να μείνω στο θέμα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται ανεξαρτήτως του ποιος παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα, γιατί αυτό έχει σημασία. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει στο εξής στοιχείο να ερμηνεύει με περιοριστικό τρόπο η Κομισιόν το άρθρο 51 και να λέει όποιες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών γίνονται μεν από τα κράτη πλην όμως αν αυτά δεν ενεργούν ή δεν εφαρμόζουν ευρωπαϊκή νομοθεσία τότε υποτίθεται δεν έχει αρμοδιότητα η Κομισιόν. Δηλαδή δημιουργείται εδώ μια γκρίζα ζώνη όπου τα κράτη θα ελέγχονται σύμφωνα με την Κομισιόν, όταν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκτελώντας ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και κατά τα άλλα, σε όλους τους άλλους τομείς θα κάνουν ό,τι γουστάρουν, θα επιβάλλουν μέτρα τα οποία είναι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα λέμε ή θα λέει η Κομισιόν ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια τέτοια ερμηνεία, ούτω ώστε να καλυφθεί πλήρως η περίπτωση της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης. Είτε από τα όργανα της Ένωσης, είτε από τα κράτη-μέλη, είτε από όργανα που κινούνται σε γκρίζα ζώνη, όπως είναι το Eurogroup. Το ξαναλέμε, το Eurogroup δεν μπορεί να είναι εκτός ελέγχου. Και φτάνουμε στην επόμενη περίπτωση που είναι τα ad hoc όργανα που λειτουργούν, όπως ήταν η Τρόικα. Διότι εδώ ήρθαμε στο σημείο να έχουμε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων εκ μέρους της Τρόικας και να απαντάει η Κομισιόν ότι δεν μπορεί να δει το θέμα διότι αυτά τα όργανα δεν είναι δίθεν όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στην πράξη είναι κάποιοι θεσμοί οι οποίοι ναι μεν μπορούν να παραβιάζουν τα δικαιώματα αλλά δεν έχει σχέση εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αποφάσεις της Τρόικας. Τα μνημόνια δηλαδή τα περίφημα. Και για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο και για την Πορτογαλία και για την Ιρλανδία. Ιδίω όμως για την Ελλάδα να υπάρχει απαγόρευση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης, να μην μπορούν δηλαδή τα συνδικάτα να διαπραγματευτούν, να μην μπορεί να γίνει συλλογική δράση και αυτά βεβαίως επιβλήθηκαν μέσα από τα μνημονιά, που ήταν παραβιάσεις δικαιωμάτων συλλογικών και μας λένε ότι δεν τρέχει τίποτε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το σημείο 7 της έκθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι επίσης στο ότι υπάρχει ήδη από 13 Μαρτίου του 2014, δηλαδή από την προηγούμενη θητεία, μια απόφαση της του Κοινοβουλίου μας για το ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας στις χώρες της Ευρωζώνης όπου εκεί έχουν παρατηρηθεί παρανομίες και ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια παρέμβαση στα ζητήματα αυτά. Και κλείνω κύριε Πρόεδρε ξαναλέγοντας αυτό που είπα πριν ότι ο κύριος Ντάισεμπλουμ ανενδίαστα σε ερώτηση που του υπέβαλα εγώ σε αυτό το σώμα εδώ στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής είπε ότι έγιναν επιλογές να διασωθούν οι τράπεζες και να επιβληθούν τα μνημόνια παρότι έτσι φτωχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός. Διότι υπάρχει ένα ερώτημα και τελειώνω. Η Ελλάδα πήρε 288 δισεκατομμύρια ευρώ με τα τρία μνημόνια. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Αν είχαν πέσει 288 δις στην Ελλάδα θα είχε απογειωθεί η οικονομία. Δεν θα ήταν κοινωνικό νεκροταφείο. Ο ίδιος ο Ντάισεμπλουμ είπε ότι έκαναν τις επιλογές για να διασώσουν τις ξένες τράπεζες και τους δανειστές. Εδώ δεν έχουμε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Πώς θα παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί λοιπόν να ισχύσουν αυτά τα οποία μας έλεγε η Κομισιόν. Και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε πρακτικά πώς θα υπάρξει αποζημίωση του ελληνικού λαού, των πολιτών, των επιχειρήσεων και του ελληνικού κράτους όπου επευλήθη ένα μνημόνιο που κατέστρεψε την οικονομία και τελικά ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, διότι τις αποφάσεις έλαβε το Eurogroup. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Äh, e. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Κούνεβα από την ΚΟΕ, e, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι σε εσά, στους συνάδελφους και στους διερμηνείς να έχουμε μια δημιουργική χρονιά μέχρι το τέλος της θητείας μας. Και ας πούμε όμως στο θέμα. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων τέθηκε σε ισχύ το 2009. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγινε προταριότητα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση από μια έννοια αγορά έγινε Ένωση Δημοκρατίας και Προστασίας των Πολιτών. Όμως αυτό ισχύει στην πράξη. Τι γίνεται με την προστασία της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, με την ιδιότητα του πολίτη και την δικαιοσύνη. Ενσωματώνεται ο χάρτης το νομοθετικό έργο μας. Έργο που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, ισότιμα με τις συνθήκες. Γνωρίζουμε από τις αναφορές που έχουν συζητηθεί, όπως ο χάρτης παραβιάζεται σε πολλά κράτη-μέλη, διότι η τήρηση του επιβάλλεται μόνο κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τι σημαίνει αυτός ο περιορισμός. Σημαίνει παράδειγμα ότι στις χώρες που επιβλήθηκαν μνημόνια και σκληρά μέτρα λιτότητας, τα μέτρα αυτά δεν είναι αναγκαίο να είναι σύμφωνα με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί υποτίθεται ότι τα μνημόνια δεν αποτελούν δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλές αναφορές που αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες είναι ανίσχυροι όταν τους επιβάλλεται αποκλεισμός από δικαιώματα όπως η συλλογική διαπραγμάτευση και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, τα δικαιώματα ψήφου, το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες, συντάξεις, το δικαίωμα σε αξιοπρεπή εργασία, και αμοιβή. Αυτά εξαιρούνται από την εφαρμογή του χάρτη στο όνομα της επικουρικότητας. Η Επιτροπή πάντα μας απαντά στις ερωτήσεις. Τι να κάνουμε, αυτό προβλέπει ο ίδιος ο χάρτης. Όμως, είναι δυνατό ο νομοθέτης που έδωσε στον χάρτη ισχύ ισότιμη με τις συνθήκες να είχε την πρόταση να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να το παραβιάσουν. Αν το άρθρο 51 του χάρτη αφήνει ανοιχτό αυτό το παράτηρο, πρέπει να το αλλάξουμε. Ακόμα και αν χρειάζεται αναθεώρηση της συνθήκης. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Τερικάμπρα για τις προτάσεις του, συμπίπτουμε στα περισσότερα. Οι τροπολογίες μας σκοπεύουν να ενισχύουν το κείμενο της γνωμοδότησής του, έτσι ώστε ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων να γίνει ισχυρό νομικό κείμενο. Οι πολίτες πρέπει να νιώθουν σίγουροι ότι έχουν ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια τους, όχι ένα ανεφαρμοστό Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Θα συνοψίσω διότι είμαι σκιώδη εισηγητής. Αλλά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, η κυρία Εύη, συγγνώμη. Μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Να ζητάτε με σαφήνεια το λόγο, να σας βλέπουμε. Okay, won't be shy. Okay. Ωραία, δεν θα ντρέπομαι. Ωραία. Λοιπόν, ε, και εγώ παρεμβαίνω εν συντομία, απλά για να πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερα τη γνωμοδότηση του εισηγητή του κ. Τερικάμπρας. Ήδη η περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι των δικών μου σκέψεων. Συμφωνώ λοιπόν και με τα όσα λέει ο εισηγητή και με τα όσα είπαν συνάδελφοι. Έχουμε μπροστά μα ε, ξαφνικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώσει επί τη αρχής ε, που πολύ συχνά ακούμε σε θεσμικό επίπεδο και που συνεχίζουν ε, να αποκρύπτουν ε, την πραγματική, το πραγματικό νόημα του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διαρκώς εισάγονται πολιτικές ε, εμπορικού χαρακτήρα περισσότερο, εξυπηρετούν τις αγορές και τη λογιστική. Οπότε πρέπει να αναστρέψουμε την κατάσταση κατά την απόψή μου. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες ε, και δύναμη όσων, είπαν και οι συνάδελφοι και ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε μια καλή συμφωνία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Πιενάρτα, από ό,τι βλέπω εδώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα ήθελα να απαντήσω στην παρατήρηση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όπως ε, γνωρίζετε, το δικαστήριο στην ε, απόφαση της 20 Σεπτεμβρίου του 2016 αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Παρότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ε, πέφτει εκτός του νομοθετικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει δεσμευμένη από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να διασφαλίζει οι δράσεις της ε, να συνανάδουν με το Χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, κατά τη σύνταξη των μνημονίων ε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας θα πρέπει να φροντίζει τα μνημόνια αυτά να ε, συμφωνούν με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό. Το δικαστήριο δεν βρήκε να υπάρχει εδώ παραβίαση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση για την οποία μιλάμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρόντισε να εφαρμοστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ακόμη λοιπόν και αν υπάρξουν άλλε επικρίσει για τα μνημόνια κατανόηση, ε, κατά τη γνώμη μα δεν υπάρχει θέμα παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικότερα όσον αφορά την ε, ερμηνεία του άρθρου 51 του χάρτη. Καταλαβαίνουμε τους ε, πολίτες που ζητάνε πιο ευρύ εφαρμογή του χάρτη, ωστόσο ο χάρτης ε, δεν μπορεί να διευρύνει τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι λοιπόν τόσο πολύ θέμα του χάρτη. Ε, έχει να κάνει με το άρθρο 6.1 της Συνθήκης της Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται λοιπόν από τις αρχές αυτές και έτσι δεν είναι δυνατόν να διευρύνουμε την εφαρμογή αυτού του άρθρου του χάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνόψησε ε, πολύ καλά το επίμαχο θέμα. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πολύ σωστά το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ό,τι έχουμε καταγράψει να εφαρμόζεται κιόλα. Ε, δίνω το λόγο τώρα στον εισηγητή και έχω μια ε, πολύ καλή είδηση για τον ε, εισηγητή. Μόλις ολοκληρώσεις την ε, παρέμβασή σου θα πρέπει να αλλάξουμε θέσεις διότι πρέπει να υποδεχθώ κάποιους επισκέπτες. Τότε πράγματι θα είσαι ο πρεσβύτερος και θα πρέπει να αναλάβεις την προεδρία. Εγώ είμαι κάπως πιο νέος. Θα ακούσουμε την παρέμβασή σου λοιπόν και μετά θα αλλάξουμε θέσεις. Μπορεί κάποιο να θεωρήσει ότι αυτό θα γίνεται κάθε φορά, αλλά όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Ναι, συμφωνώ, είναι δύσκολο για την Επιτροπή, αλλά αφού η γλώσσα είναι τόσο σημαντική, είπατε ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή. Η Κομισιόν όμως και όλοι μας μπορούμε να επεκτείνουμε την ερμηνεία διότι το εφαρμόζουμε μετά από ερμηνεία, βάση ερμηνεία. Εάν ερμηνεύσουμε κάποιε αρχέ ή κάποιου όρου με έναν τρόπο, τότε τι εφαρμόζουμε με τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο. Αλλά ξέρω, ναι, υπάρχουν κάποιε δυσκολίε ε, και όπω είπε και ο πρόεδρο, είμαστε σε επαφή με την ΑΦΚΟ και πρέπει να το ενισχύσουμε το κείμενο έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον επαφών. Ευχαριστώ όμως και τους συναδέλφους. Νομίζω ότι συμφωνούμε επί πολλών. Ε, σημείων. Τόσο που πιστεύω με τις τροπολογίες η γνωμοδότηση θα είναι πολύ ικανοποιητική. Αυτό ελπίζω και εύχομαι. Ευχαριστώ. Και ε, ως ανταμοιβή για τις εργασίες σου θα αναλάβεις την Προεδρία της Επιτροπής. Παρακαλώ. Finally I got power. Finally. Ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους ε, ε, έφτασα στην εξουσία. Είναι κάτι για το οποίο αγωνίζομαι επί μήνες και χρόνια. Επιτέλους λοιπόν. Θέλετε να πάρετε το λόγο πριν ξεκινήσουμε. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στην ε, γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό υπαριθμών 1 κάθετος 2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια είναι η αγαπητή φίλη η κυρία Βαλίνα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μετά την συζήτηση που είχαμε τον Ιούλιο στην Επιτροπή μας, για διάφορες αναφορές που έχουν να κάνουν με την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να αρχίσω ευχαριστώντας τους αναφέροντες για την προσπάθεια που κάνουν. Εγώ λοιπόν παρουσιάζω αυτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, που είναι γνωμοδότηση στην Επιτροπή Γεωργίας, που είναι η αρμόδια επί της ουσίας θέλω να τους ζητήσω, εννοείται, να λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις μας, τις προτάσεις μου. Στην γνωμοδότησή μου, λοιπόν, υπογραμμίζω πρώτα απ' όλα ότι η Επιτροπή Αναφερών έχει, αν, έχει παρελάβει πάρα πολλές αναφορές, πολυάριθμες, που καταγγέλουν ε, την μεταφορά των ζώων. Ε, παραβιάζονται συστηματικά οι κανόνες και δεν τηρούνται οι κανονισμοί ούτε από τις χώρες μέλη, ούτε και από τους ίδιους τους μεταφορείς. Γι' αυτό και καταδικάζω και εγώ αυτήν την κατάσταση και λέω ότι δεν είναι δυνατόν 13 χρόνια αφότου άρχισε να ισχύει ο κανονισμός να εξακολουθούν να μεταφέρονται ζώα κάτω από συνθήκε που είναι πραγματικά τραγικές. Στη γνωμοδότηση αυτή λοιπόν ζητώ από όλε τις χώρες μέλη να φροντίσουν τα ταξίδια, μεταφορά των ζώων να προγραμματίζεται από την αρχή μέχρι το τέλος της μεταφοράς βάση των κανόνων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταφορά των ζώων, να λάβουν υπόψη τους ακραία καιρικά φαινόμενα, να λάβουν υπόψη τους ε, τον τρόπο μεταφοράς, το μέσο μεταφοράς και τις ε, γεωγραφικές ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός. Και επαναλαμβάνω και την έκκλησή μου, ο χρόνο μεταφοράς των ζώων που πάνε στα σφαγεία να περιορίζεται στις 8 ώρες, λαμβάνοντας υπόψη υπόψη βέβαια και το χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης, αλλά και το διάστημα που περνούν στα σύνορα για τους ελέγχους στα φορτηγά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που συνδέονται με τα τεράστια, το τεράστιο χρόνο μεταφοράς των ζών θα λυνόταν αν τελικά η μεταφορά δεν γινόταν μεταφορά ζών αλλά μεταφορά του κρέατος μόνο. Οπότε, ο κανονισμό δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο. Πολλέ χώρε δεν ελέγχουν, δεν προβαίνουν σε ελέγχου και δεν φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων. Και κάποιοι μεταφορεί επίση να ξέρετε ότι δρούν παράνομα. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομένου ότι δεν υπάρχει αναρμόνιση στου ελέγχου και στι κυρώσει στι χώρε μέλη να σκεφτεί τη δυνατότητα αναθεώρησης των σημερινών διατάξεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ισχύουν τα ίδια, οι ίδιοι μηχανισμοί κυρώσεων δηλαδή, σε όλες τις χώρες, που να είναι εξίσου αποτελεσματικοί. Καταδικάζω επίσης το γεγονός ότι δεν τηρείται ο κανονισμός ε, σχεδόν καθόλου όταν πρόκειται για τη μεταφορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ζητά από τους μεταφορείς να τηρούν τους κανόνες σε όλη τη διαδρομική εκείνη που λαμβάνει η χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες μέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να έχουν συνεπή συστήματα επίσης ε, συλλογής στοιχείων και για τα ζώα τα άρρωστα ή τα πληγωμένα που πηγαίνουν σε τρίτες χώρες και να φροντίζουν να γίνονται οι επιθεωρήσεις που πρέπει. Τέλος, δεδομένων αυτών των συστηματικών προβλημάτων τήρησης των κανόνων, να φροντίσει για τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες μέλη. Να αρχίσουν αμέσως οι έρευνες που χρειάζονται για να δούμε τι παραβιάσεις έχουν γίνει στους κανονισμούς και βεβαίως να ξεκινήσει ε, διαδικασίες κατά παραβάση σε βάρος των υπεύθυνων χωρών. Τίποτα άλλο, είμαι στην διάθεση των σχεδόν εισηγητών εννοείται για να συνεργαστούμε με τις άλλες πολιτικές ομάδες δηλαδή για να μπορέσει η Επιτροπή μας με την γνωμοδότηση αυτή να βελτιώσει τις πρακτικές και την τήρηση των κανονισμών. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Προσγέρη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά διότι μιλώ εκ μέρου τη Μέλεν Μίτζη, Η κυρία Μίτση θα ήθελα να ζητήσει συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεση για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία είναι σκιώδη. Καλωσορίζει τη γνωμοδότηση τη κυρία Βαλίνα για τι μεταφορέ εντό και εκτό Ευρώπη και υποστηρίζει του γενικού στόχου. Η γνωμοδότηση εστιάζεται στη σπουδαιότητα των αναφορών που υποβάλλουν οι πολίτε για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά που συχνά καταγγέλουν συστηματικέ συνεχεί και σοβαρέ παραβιάσει του κανονισμού 1-2005 από τα κράτη-μέλη και από του μεταφορεί. Η κυρία Μίτση συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι είναι απαράδεκτο 13 χρόνια μετά από τη θέση ισχύ του κανονισμού ακόμα να μεταφέρονται ζώα στι φρικιαστικότερε συνθήκε, κατά παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού 1 2005 θα πρέπει να εφαρμοστεί η υπάρχουσα νομοθεσία καλύπτοντα όλα τα ζώα ανεξάρτητα από τον τρόπο ανεξάρτητα από τι συνθήκε εντό χερσαίο ή θαλάσσιο, ανεξάρτητα από τι συνθηκε εντο ή εκτο τη Ευρω... της Ευρωπαϊκής Η κυρία Μίτση επιση υποστηρίζει την προσέγγιση τη εισηγητρία για να υπάρξει ένα σύστημα παρακολούθηση τη συμμόρφωσης με τον κανονισμό σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να ξεκινούν ε, έρευνες πιθανών παραβιάσεων του κανονισμού και να ε, ξεκινούν ε, διαδικασίες κατά παραβάση κατά των αρμόδιων κρατών μελών. Θα κάνει και ποια προσθήκη η κυρία Μίτση στο κείμενο δεδομένων αυτών. Πιστεύει ότι αυτή θα συμβάλλει θετικά στο καλό πνεύμα του σχεδίου γνωμοδότησης, στέλνοντας ένα ικανοποιητικό μήνυμα προς τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη για να σταματήσει η κακή μεταχείριση των ζώων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανε η συγγήτρια, η κυρία Βαλίνα και να πω ότι μια και λύσαμε το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τώρα ερχόμαστε στην προστασία των δικαιωμάτων των ζώων. Εδώ λοιπόν δεν θα γίνει διαφοροποίηση. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν παραβιάζουν τα δικαιώματα των ζώων ή όχι. Διότι προηγουμένως συζητούσαμε ότι τα κράτη-μέλη όταν δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν και δεν ελέγχονται από την Κομισιόν για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα τα κράτη-μέλη θα παραβιάζουν ή παραβιάζουν τα δικαιώματα των ζώων χωρίς να κάνουμε διαφοροποίηση εδώ. Για να δείξω τον παραλογισμό που υπάρχει και όχι βεβαίως να αμφισβητήσω το δικαίωμα, μάλλον τον έλεγχο που πρέπει να γίνει στα κράτη-μέλη για την παραβίαση των δικαιωμάτων των ζώων. Μια μικρή παρατήρηση στην Κομισιόν έφυγε. Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρθηκε αφορούσε κρίση για το μνημόνιο πριν ομολογήσει ο Ντάισεμπλουμ ότι όσα έκανε το Eurogroup ήταν για να σώσει τις τράπεζες και όχι τον ελληνικό λαό. Έρχομαι λοιπόν εδώ στην παρατήρηση και στην εισήγηση που έχουμε μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένο ότι υπάρχει καραμπινάτη παραβίαση των δικαιωμάτων των ζώων όπως προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεύτερον, είχαμε πάρα πολλές αναφορές στο ζήτημα αυτό. Τρίτον, είναι δεδομένο ότι η παραβίαση και η κακομεταχείριση των ζώων επηρεάζει όχι μόνο την υγεία τον ίδιο των ζώων αλλά και των ανθρώπων. Διότι αυτά τα ζώα οδηγούνται στην αγορά και στην κατανάλωση. Τέταρτη παρατήρηση έχει σχέση με το χρόνο που αφιερώνεται στη μεταφορά των ζώων. Και εδώ αυτό πρέπει να το δούμε διότι υπάρχει πολλές φορές αργοπορία λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων σε σχέση με τη μεταφορά των ζώων είτε από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Πρέπει να υπάρξει βεβαίως συμμόρφωση των μεταφορέων και επίσης συμμόρφωση σε σχέση με τα δρομολόγια. Και επιπλέον πρέπει να ληφθούν μέτρα και από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν διότι γίνονται παράνομες ελληνοποιήσεις ζώων Έχουμε δηλαδή εισαγωγές ζώων από τα Σκόπια και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία τα οποία εμφανίζονται δίθεν ως ελληνικά. Και αυτό γίνεται πολλές φορές το Πάσχα όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση αμνοερυφίων. Να υπάρξει λοιπόν αποφασιστικός έλεγχος στο θέμα αυτό για να μπορούμε από εκεί και πέρα να έχουμε ένα συνολικό πακέτο προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων ελπίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα πλήρε πακέτο προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων, δηλαδή των πολιτών τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Herr Weitz. Βάιτς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ και η πολιτική μου ομάδα έχουμε διαφορετική θέση σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει η γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη και πιστεύω ότι αυτό είναι γενικά γνωστό. Ε, αλλά το θέμα εδώ είναι οι κανόνες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταφορά ζώων να εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, από ε, την Στηρία είδαμε μεταφορά με ε, πολύ κακές συνθήκες για τα ζώα. Είχαν κρεμάσει τα ζώα, τα είχαν δέσει από το λαιμό. Ε, από την γιατρικής ε, άποψη αυτό είναι πρόβλημα, όπως και όσον αφορά την ανθρώπινη ιατρική. Επίσης, ε, όσον αφορά τους ελέγχους στο πέρασμα του Μπρένερ, και δεν πραγματοποιούνται οι έλεγχοι. Για παράδειγμα, τα νέζικο ε, όταν ε, είχε σταματήσει ήδη άκουσα τους χείρους μέσα να διαμαρτύρονται και μάλιστα ένας ήδη είχε πεθάνει. Ναι, μπορεί τα πράγματα να είναι κάπως καλύτερα στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά τέλεια δεν είναι. Πολλοί από τους ε, ιατρούς ελεγκτές δεν γνωρίζουν τους κανόνες και έτσι δεν μπορούν να ελέγξουν αν εφαρμόζονται σωστά σε άλλο έλεγχο, στην ε, Κροατία. Ε, είδα την ε, φόρτωση 4.000 βοηδών σε πλοίο. 36 βαθμοί η θερμοκρασία στο πλοίο, στα φορτηγά πάνω από 50 βαθμούς. Ε, τα ζώα δεν μπορούσαν να σταθούν όρθια διότι είχαν αφυδατωθεί. Ε, το πλοίο αυτό πήγαινε στο Λίβανο παρεπιπτόντος. Θα μπορούσα να σας δώσω και άλλα παραδείγματα ε, από τα βουλγαρικά σύνορα όπου τα φορτηγά περιμένουν επί ώρες ενώ θα πρέπει να δείτε δίνεται προτεραιότητα στις μεταφορές ζώων. Ε, μερικές φορές ε, πηγαίνουν τελικά σε άλλο μέρος σε δίθεν για ε, εκφόρτωση, αλλά που δεν γίνεται τελικά. Επί καμιά ώρα θα μπορούσα να συνεχίσω να σας δίνω πληροφορίες σχετικά με αυτά που έχω δει με τα δικά μου μάτια. Το θέμα είναι, σκεφτείτε, 120 φορτηγά από την Ιρλανδία στην Κροατία, από τη Γαλλία, από την Σλοβακία, από τη Γερμανία, από όλη την Ευρώπη. Ούτε ένα φορτηγό δεν ε, ελέγχθηκε, ενώ η αστυνομία ήταν παρούσα. Ε, κανονικά η αστυνομία δεν κάνει τους ελέγχους. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα μία άνευ προηγουμένου αποτυχία του συστήματος ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή, όχι μόνο από ευγένεια, αλλά από βαθιά πεποίθηση. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ε, και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν στηρίζουν αυτού του είδους τη μεταχείριση των ζώων και ζητούν επιγόντως να γίνει κάτι για το θέμα αυτό. Ως ε, σκιώδης ε, εισηγητής θα εργαστώ σε τούτη την Επιτροπή, θα είμαι όμως σκιώδης εισηγητής και στην άγκρη του, της πολιτικής ομάδας των Πρασίνων. Θέλουμε λοιπόν να οξύνουμε τους κανόνες, όχι να τους κάνουμε πιο χαλαρούς. Όπως σας είπα, είναι έτοιμα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών της Ευρώπης να τηρούνται οι κανόνες, ακόμα και αν θεωρούμε ότι αυτοί οι κανόνες δεν είναι αρκετά σαφείς και είναι υπερβολικά χαλαροί. Τουλάχιστον όμως ε, αυτά που έχουμε θεσπίσει να τα εφαρμόζουμε. Σας ευχαριστώ. Äh, Αυτά που μας είπατε είναι πράγματι πολύ σκληρά και απαράδεκτα. Η συνάδελφος Εύη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σκιώδη συγκήτρια για αυτή τη σημαντική έκθεση ήθελα να παρέμβω. Πρώτα απ' όλα για να εκφράσω το πόσο καλή δουλειά ήταν η δουλειά της συναδέλφου Βαλίνα σε αυτό το πρώτο σχέδιο αυτής της γνωμοδότησης που θα πάει στην Επιτροπή Γεωργίας. Ε, είναι μια εξαιρετική αφετηρία. Θα πρέπει να ενδυναμωθεί σε πολλές πτυχές. Πτυχές κυρίως ε, που αφορούν λεπτομέρειες. Έχουμε εκατοντάδες πληροφορίες, καταγγελίες, αναφορές για το θέμα αυτό και παντού βλέπουμε αυτό το θέμα που ανέφερε και ο συνάδελφος ε, με τρόπο πολύ ακριβή. Βρισκόμαστε ενώπιον ε, καταστάσεων εξωφρενικών, απαράδεκτων πλέον και που παραβιάζουν σταθερά τους κανόνες που σήμερα έχει θεσπίσει η Ευρώπη. Αυτό είναι το ζήτημα το σημαντικό. Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει και μας απαντά. Έχει απαντήσει σε πολλούς βουλευτές και σε μένα μεταξύ άλλων, σε διάφορες επιστολές που έχουμε στείλει όλους τους τελευταίους μήνες ζητώντας εξηγήσει, μεγαλύτερη προσοχή, περισσότερους ελέγχους. Περισσότερη προσοχή στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο Επίτροπος Ανδριοκαϊτής μας απαντά ότι η συμμόρφωση όσον αφορά τον κανονισμό για τις μεταφορές τον 1 του 2005 που συζητάμε και εδώ είναι σχεδόν 100% η συμμόρφωση. Παρότι εκ των πραγμάτων ούτε υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία και δεδομένα όσον αφορά τα ταξίδια που γίνονται, τις διαδρομές που γίνονται. Δεν έχουμε δηλαδή μια σαφή απεικόνηση της σημερινής κατάστασης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς είναι δυνατόν να μας απαντά κάτι τέτοιο η Κομισιόν. Το θεωρώ απαράδεκτο να αρνείται η Κομισιόν την ύπαρξη του προβλήματος. Επίσης να θυμίσω ότι η έκθεση αυτή ε, είναι μεν πολύ σημαντική αλλά δεν πρέπει να φυσικάζουμε. Ε, έχουμε ζητήσει εμεί μια επιτροπή εξεταστική ειδικά για αυτό το σημείο. Θα πρέπει να το ζητήσουμε και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες για αυτό, διότι για μένα παραβιάζει όλο αυτό τι δημοκρατικές αρχές, αρχές αυτού του θεσμικού οργάνου. Θα έπρεπε να ψηφιστεί αυτό το να υπάρξει μια εξεταστική επιτροπή. Δεν έγινε όμως. Ε, έχουμε τώρα την έκθεση. Ελπίζω να μπορέσουμε εμεί ω Επιτροπή να συμβάλλουμε με τον πιο φιλόδοξο και ε, ισχυρό τρόπο για την προστασία των ζώων, διότι δεν βλέπω να γίνεται το ίδιο πράγμα από άλλε επιτροπέ του Κοινοβουλίου και ειδικότερα από την Επιτροπή Γεωργία, που όπω γνωρίζουμε όλοι χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες ε, επιτροπές. Σας εύχομαι λοιπόν καλή δουλειά και από τη δική μου άποψη εγώ θα υποβάλω πολλές ε, τροπολογίες ε, για να αναφέρουμε και να τεκμηριώσουμε τις πολλές παραβιάσεις που βλέπουμε καθημερινά και που αξίζουν την προσοχή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η Κομισιόν. Ο κύριος Τέρνς Κέσεβι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι παρακολουθούμε προσεκτικά τα τελευταία χρόνια τις εξαγωγές ζώων των ε, ζώων. Είναι ένας ε, αυξανόμενος τομέας του εμπορίου και έχουμε πολλά στοιχεία για το θέμα αυτό. Λέτε ότι πρόκειται για μικρό ποσοστό, αλλά επειδή μιλάμε για μεγάλο όγκο, μπορεί και πάλι να μιλάμε για μεγάλο αριθμό μεταφορών. Το βασικό πρόβλημα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και είναι κάτι το οποίο επισήμανε σε όλους τους συναδέλφους του ο Επίτροπός μας ε, φέτος. Επίσης όλες οι αρχές ε, έχουν ε, ενημερωθεί. Το βασικό μέτρο που μπορεί να ληφθεί στις περιπτώσεις αυτές είναι να σταματήσει η μεταφορά. Ε, αυτή είναι πολύ σημαντική κύρωση, διότι απαιτεί πολλή προετοιμασία μια τέτοια μεταφορά. Αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές και έχουμε ακούσει παρατηρήσεις των αρμοδίων αρχών. Εξετάζουμε λοιπόν ποιες μεταφορές δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη συμμόρφωσης. Ωστόσο βλέπουμε ότι κάποιες μεταφορές πραγματοποιούνται παρά τις προειδοποιήσεις ε, του Επιτρόπου. Ε, ιδιαίτερα στα τουρκικά σύνορα έχουμε δει προβλήματα και οι αρμόδιες αρχές ε, γνωρίζουν το πρόβλημα. Συνεχίζονται οι έρευνες και βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και με τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους σε σχετική κατάρτιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαλίνα έχει τη δυνατότητα... Θέλετε να μιλήσετε? Just one word for the commission. Δύο λόγια απλά για την Κομισιόν. Ξέρετε κάτι, υποτιμάτε το πρόβλημα. Ναι, η θερμοκρασία είναι ένα πρόβλημα και ο τεχνικός εξοπλισμός και τα χρονικά πλαίσια είναι πρόβλημα. Οι μεταφορείς κλέβουν, σας κοροϊδεύουν περιγράφουν ε, σημεία εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των ζώων και τα αναφέρουν ως προορισμούς των ζώων παράνομα. Ένα σωρό παρανομίες γίνονται. Τα ξέρετε στην Κομισιόν και στο τμήμα σας. Μην υποτιμάτε τη σοβαρότητα του προβλήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βαλίνα θέλει το λόγο voy a hacerlo más Θα είμαι σύντομη, γιατί πράγματι τα είπε ο συνάδελφο όλα όσα σκόπευα να πω. Όντω, δεν φτάνουν όλα αυτά. Είναι ανεπαρκή αυτά που κάνετε. Βλέπω πάντως ότι είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή. Και ως συντάκτρια της γνωμοδότησης, έχω περιορισμούς βέβαια στην έκταση της γνωμοδότησης, αλλά αφού είμαστε στην ίδια γραμμή, ε, ευχαρίστως να βελτιωθεί με τις τροπολογίες των συναδέρφων για να γίνει έτσι όπως όλοι θέλουμε. Ό,τι μπορείτε να βελτιώσετε στη γνωμοδότηση αυτή είναι ευπρόσδεκτο. Οι περιορισμοί είναι αυτοί που ξέρουμε, οπότε οι συνάδελφοι μπορούν να εμπλουτίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να σας θυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 6η Σεπτεμβρίου, δηλαδή η 5η υποβάλλεται παρακαλώ μέχρι τις 3 ε, ε, το μεσημέρι. Οπότε υποβάλλεται ε, τροπολογίες ε, καλές και που να κάνουν κάποια αλλαγή. Πρόεδρε, πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ήθελα να κάνω μια δήλωση. Έμαθα ότι η ο εισηγητής για τη μεταρρύθμιση του εργαλείου ε, πρωτοβουλία των πολιτών δεν παρετείται από αυτό το αρχείο. Δεν θα είναι αυτός που θα κάνει το αρχείο αυτό. Και ήθελα απλά να πω εδώ ότι θεωρώ ότι δεν είναι σωστό ότι ανατίθεται ξαφνικά στα γρήγορα το θέμα αυτό και ότι αναβάλλεται ε, το ζήτημα αυτό για συζήτηση στους συντονιστές διότι τότε οι συντονιστές ε, είχαμε μείνει ικανοποιημένοι με το να συνεχίσει ο Βαλένσα ως εισηγητής αυτού του αρχείου όπως και γίνει με την ε, έκθεση πρωτοβουλίας που είχε προηγηθεί αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των συντονιστών και όχι όπως έγινε αυτή τη στιγμή το ότι δόθηκε προτεραιότητα όσον αφορά τις πολιτικές ομάδες και βάσει αυτής έγινε η ανάθεση θεωρώ ότι θα έπρεπε να ξανασυζητηθεί στους συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ. Το σημειώνω τα όσα είπατε. Συμφωνώ κιόλα. Θα το συζητήσουμε στις 24 του μήνα στη συνάντηση των συντονιστών. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ και προσπαθήστε να μείνετε ευτυχείς.